Okay, colleagues, may have your attention, please. Συνάδελφοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Ο κύριος Στόγερ έρχεται. Θα είναι εδώ σε 15 λεπτά. Προτείνει όμως να ξεκινήσουμε το μεταξύ. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την οποία λάβετε στις 26 Σεπτεμβρίου και βρίσκεται και στο φάκελο που έχετε για αυτή τη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας μιλήσω ε, για το γλωσσικό καθεστώς. Ε, το οποίο γνωρίζετε. Βρίσκεται ένα χαρτί στο φάκελο με τα έγγραφα της συνεδρίασης. Ε, υπάρχει ε, δημόσια εκπομπή για αυτή τη συνεδρίαση. Να σας πω επίσης ότι πρέπει να υπογράψετε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν φύγουμε για το Λουξεμβούργο. Για το Λουξεμβούργο. Έγιναν κάποιες αλλαγές στη γραμματεία ε, δύο συνάδελφοι έφυγαν από τη γραμματεία και ο κύριος Πίνταλ έρχεται. Ε, σας ε, συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εάν όμως ο η, εισηγητή, η θέλει να πει κάτι, ε, έχετε το λόγο. Κύριε Γκρέσλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Έστειλε σε όλους τους αδέλφους ένα mail μετά την τελευταία αναβολή όπου προσπάθησα να εξηγήσω την κατάσταση και νομίζω ότι μπόρεσα να άρω ε, όλες τις ανησυχίες όσον αφορά την άρση ασυλία των μελών. Γνωρίζετε ότι το αίτημα το οποίο ήρθε καθυστερημένα δεν κρίτη από το Συμβούλιο. Στην αρχή υπήρχε κάποια προθυμία προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλοι όσοι παρίσταντο γνωρίζουν ότι ε, το προσπάθησα και δεν το κατόρτωσα και συμφωνήσαμε τελικά η Κομισιόν να προβεί σε δήλωση, ίσως ο Επίτροπος κύριος Σεμέτα και χαίρομαι που βρίσκεται εδώ να τοποθετηθεί από αυτού, να μας πει τι θα γίνει με αυτή τη δήλωση και θέλω να πω ότι αν πρέπει κανείς να επεξεργαστεί το θέμα της άρσης ηλίας μελών, τότε θα πρέπει να γίνει με βάση το καταστατικό των βουλευτών. Δηλαδή ε, αυτό με τα άρθρα δεν ε, ήταν αποτελεσματικό. Το προσπαθήσαμε αλλά δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Και παρεπιπτόντως αυτή η τροπολογία η οποία δεν έφτασε ποτέ στην Ολομέλεια ε, το να αποτύχουν τα πάντα λόγω αυτής της τροπολογίας θα ήταν κρίμα. Κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί ποτέ δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά στην τροποποίηση της Όλαφ όπως έχουμε φτάσει τώρα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για όλους μας το γεγονός ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και ελπίζω να δεχτείτε όλοι σας το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμμετείχαν, όλους όσοι παρέμειναν στην τριμερή συνάντηση. Να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου, την Πολωνική Προεδρία και κυρίως την Προεδρία της Δανίας που έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά η Ουγγρική Προεδρία έκανε την αρχή και γι' αυτό θέλω να πω ότι θα ήταν πραγματικά κρίμα και πολιτικά ανόητο εάν δίναμε την εντύπωση στα κράτη-μέλη ότι φταίμε εμείς, ότι εμείς οδηγήσαμε στην αποτυχία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχετε μπροστά σας είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα γιατί για πρώτη φορά μας δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί το θέμα της αντιμετώπισης απατών. Και είμαι σίγουρη ότι αν το συζητήσουμε το θέμα αυτό από κοινού με την Προεδρία, με την Όλαφ, με την Επιτροπή, με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα και θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία στην καταπολέμηση των απατών από ό,τι μέχρι τώρα. Εγώ ένα πράγμα βρίσκω πολύ δύσκολο. Να λένε όλοι, ε, σημαντικό το θέμα, ε, το λέμε καθημερινά, αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα κανείς δεν κάνει τίποτα. Η κατάσταση λοιπόν τώρα άλλαξε και πραγματικά μεριμνούμε έτσι ώστε στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα να προχωρήσουμε καλύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ευχαριστώ θερμά την μικρή ομάδα εργασία, την συνεργατητά μου, την κυρία Φραντσέλο, την νομική υπηρεσία, την κυρία Ντεμπράτσκα, ε, τους δύο νομομαθείς, ε, γλωσσομαθείς νομικούς, Τις δύο κυρίες μάλλον είναι οι οποίες μας βοήθησαν πάρα πολύ, την κυρία Ρατσόνη, την κυρία Ούλριχ, την προκάτοχό της. Ευχαριστώ όλους αυτούς ε, θερμά. Ευχαριστώ θερμότατα τους ε, συναδέλφους και τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων που συνέβαλαν. Γιατί όλοι συνέβαλαν στο να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας ανέφερα. Προτείνω λοιπόν ο κύριος Επίτροπος να τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις τη Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια σχόλια πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Ε, τότε, κύριε Στές, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι με ικανοποιεί απολύτως η δουλειά της κυρίας Γκρέσλε άνευ προηγουμένου είναι αυτό το οποίο έχει γίνει, δηλαδή να έχει προσεγγίσει ένα φάκελο με τέτοιο τρόπο. Ε, την περασμένη φορά που συνεδριάσαμε καταλήξαμε σε κοινή συμφωνία και θα ήθελα να δηλώσω πόσο καλή βούληση θέλουμε να δείξουμε ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητες και θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους συνεδριάσεις και μάλιστα εγκαίρως για να μπορέσουμε να συμφωνούμε ε, με πιο, σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα και αρκετά εγκαίρως, όχι όπως αυτή τη φορά. Να ευχαριστήσω πάλι όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στά, συγγνώμη, ε, ο κύριος Επίτροπος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα σκοπό να μιλήσω εκτεταμένα στην επόμενη μου παρέμβαση, όταν θα σχολιάσω τις, πρωτοβουλίε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα καταπολέμησης της απάτης. Θα έχω την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσω και αργότερα. Προς το παρόν, ε, σε αυτό το στάδιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε και όλους ε, όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα. Πράγματι, χρειαστήκαμε πολλά χρόνια εγώ μέτρησα έξι, η κυρία Γκρέσλε μέτρησε 8. Μπορεί και να είναι 8. Χρειαστήκαμε πολλά χρόνια, αλλά έχουμε φτάσει σε μια καλή συμβιβαστική λύση, η οποία θα εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης, η Όλαφ, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και θα κινείται σε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο πλαίσιο στις δραστηριότητες της στο μέλλον. Ε, υπήρξαν ε, ζητήματα αντιφατικά και η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε δύο δηλώσεις με την έγκριση του κανονισμού. Η πρώτη θα έχει να κάνει με τις εργασιακές ρυθμίσεις ε, ανάμεσα στην Όλαφ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εκεί θα διευκρινίσουμε ξεκάθαρα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων μερών. Η δεύτερη δήλωση της Επιτροπής θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο για τις ασυλίες και για ε, τον εσωτερικό κανονισμό των μελών. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν θα προσαρτηθούν στον κανονισμό και νομίζω ότι με αυτές τις δηλώσεις θα καταλαγιαστούν όλες οι ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κανονισμό αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρατηρήσεις προτείνω να προχωρήσουμε. Κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω την Όλαφ και τον Γενικό της Διευθυντή. Καλώς. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Ας προχωρήσουμε με την ψηφοφορία για την ενδιάμεση έκθεση για τον κανονισμό του Συμβουλίου που καθορίζει ε, το νέο πολιτές με δημοσιονομικό πλαίσιο. Α, να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ενδιάμεση έκθεση ή για την Όλαφ. Με συγχωρείτε, διακόπτη η Προεδρεύουσα. Είναι μια ψηφοφορία ναι ή όχι. Ποιος είναι υπέρ. Να σηκώσει το χέρι του. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Οκ. Okay. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Τώρα λοιπόν πάμε, μετά που ψηφίσαμε στην ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Η συγητής είναι ο κύριος Μάλντερ. Θα ήθελα να ε, ζητήσω ε, ε, να μάθω ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 1. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Επόμενο σημείο. Στην ημερήσια διάταξη. σχέδιο έκθεσης για την πρόταση κανονισμού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που θα καθορίζει τους κανόνες για τις άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθα καθεστώτων στήριξη τη κοινή γεωργική πολιτική. Συντάκτρια γνωμοδότηση η κυρία Χολμάιερ. Τροπολογία 20. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού για την 20. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Πάλι ηλεκτρονικά προτείνω να ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για της ηλεκτρονικής οδού. Για την 57. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 αποσύρεται. 25 αποσύρεται. 26 και 27 το ίδιο. 63, 63 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62. Καταπιπτεί 62 εάν η 63 εγκριθεί όπερ και αγένετο. Τροπολογία 28. Λοιπόν, αυτές οι τρεις καταπίπτουν, οι 28, 29 και 30. Την 64 ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, υπέρ. Κατά, αποχές, δεν ήταν καθόλου σαφές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 31. Ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 και 33 έχουν αποσυρθεί. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 Υπέρ. Κατά. Δεν ήταν σαφές να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 67. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 39 αποσύρεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 αποσύρεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 42 αποσύρεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 43 έχει αποσυρθεί. Η 44 μαζί με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 και 46 και 47 και 48 είναι τροπολογίες που αποσύρονται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 και 51 αποσύρονται. 53 ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 αποσύρεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγ... απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 6 αποσύρεται, 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 9 και 10 αποσύρονται, 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 12 έχει αποσυρθεί, 13. Σε τρία τμήματα όπως το βλέπω ή σε δύο, σε δύο μάλλον τμήματα. Πρώτο τμήμα της 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν ήταν σαφές, ψηφίζουμε για τις ηλεκτρονική οδού το πρώτο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 13. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14, 15, 16. Αποσύρονται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία δια της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κύριε Γκάιερ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, είχα το εξής πρόβλημα, ότι στο γερμανικό κανάλι παρισέφρισαν και άλλες γλώσσες και αυτό με αναστάτωσε, μου προκάλεσε σύγχυση. Γι' αυτό λοιπόν εκεί όπου ψηφίσαμε για την τροπολογία 58 του κυρίου Σκυλακάκη ε, στην πρώτη σελίδα, τη στιγμή που εσείς ε, αναφέρατε αυτή την ε, τροπολογία, για τους λόγους που σας εξήγησα, τα πράγματα ήταν μπερδεμένα και εγώ δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Απορρίφθηκε η τροπολογία λόγω του 20 αυτό ήταν το αποτέλεσμα, ψηφία. Εγώ θέλω να υπερψηφίσω και θα εγκριθεί η τροπολογία. Παρακαλώ να το καταγράψετε στα πρακτικά. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα λάβουμε υπόψη μας την παρατήρησή σας. Κύριε Γκρέσλα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που είπατε, αλλά αυτό δεν ξέρω. Πρώτη φορά επιτρέπεται εκ των υστέρων να αλλάξει το αποτέλεσμα μιας ε, ψηφοφορίας. Ε. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι στον κανονισμό κατά πόσον είναι δυνατόν να αλλάξει εκ των υστέρων αποτέλεσμα τροπολογίας και ψηφοφορίας κυρίως. Ευχαριστώ. Σημείο 6. Απαλλαγή 2011 τμήμα 3, Επιτροπή. Έχουμε τον Επίτροπο κύριο Σέμετα σήμερα μαζί μας. Να του δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω διότι σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και ενδιαφέρει ιδιαίτερο στη δική σας Επιτροπή. Καταρχάς, η έκθεση παρακολούθησης. Σε αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει με πολλές λεπτομέρειες τα μέτρα και τα τις δράσεις που έχουν αναλυφθεί κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κατά τη διαδικασία της απαλλαγής του 2010. Δεύτερον, η συνθετική έκθεση, η έκθεση σύνθεσης για το 2011, είναι μια έκθεση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την πολιτική της ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων και την επίτευξη των στόχων. Και τέλος, έχουμε την ετήσια έκθεση για τους εσωτερικούς ελέγχους, η οποία διενεργήθηκε το 2011. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον εντοπισμό των τάσεων ε, στη διαχείριση των προϋπολογισμών. Θέλετε να δείτε εάν οι δράσεις που αναλήφθηκαν βάσει συστάσεων πράγματι κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση. Το ίδιο επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ε, να συγκρίνουμε την απόδοση, την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προπολογισμού και μας βοηθά να εντοπίσουμε και τα αδύναμα σημεία στα οποία πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την έκθεση παρακολούθησης. Έχετε λάβει τρία έγγραφα. Μια σύντομη έκθεση που παρουσιάζει την παρακολούθηση ε, βάσει των πιο κρίσιμων ετοιμάτων του Κοινοβουλίου, τις τέσσερις δράσεις προτεραιότητας από τη μία και τα βασικά αιτήματα που έχουν να κάνουν με τους κύριους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Έγγραφα εργασίας ε, περιλαμβάνουν τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε μία ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, των συστάσεων του Συμβουλίου. Ας μιλήσουμε για τις, ε, τέσσερις δράσεις προτεραιότητας που έχουμε συζητήσει εκτενώς με εσάς πριν από την ψηφοφορία το Μάιο. Πρώτη δράση προτεραιότητας, πιο στενή παρακολούθηση της χρήσης των ε, ε μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Ετροποποιήσαμε το υφιστάμενο ε, νομοθετικό πλαίσιο και θα κάνουμε ε, παρουσίαση έκθεσης προς την αρχή που δίνει την απαλλαγή. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν με χαρά μου σας ενημερώνω ότι μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα θα λάβετε λεπτομερή έκθεση για το πώς τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υφίστανται αυτή τη στιγμή, πώς θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται και πολλές από τις αιτήσει, από τα αιτήματα ε, υπό τη δράση προτεραιότητας 2, δηλαδή βελτίωση της αλυσίδας λογοδοσίας της Επιτροπής. Θα θυμάστε ότι στη δική σας Επιτροπή έχω υποβάλει όλες τις αιτήσει περιλήψεις και εκθέσεις για όλα τα κράτη-μέλη και θα συνεχίσω να το κάνω διότι σέβομαι πλήρως το ρόλο της αρχής που δίνει την απαλλαγή για τον προπολογισμό βάσει της συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βελτιώσει ετή περαιτέρω την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των εκθέσεών μας. Ε, οριζόντια σε όλες τις υπηρεσίες μας έχουμε δώσει εντολές που λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για να ε, απαντήσουμε στα αιτήματα της Επιτροπής σας, δηλαδή πώς θα υπολογίσουμε το ποσοστό σφάλματος, πώς θα υπολογίσουμε τους κινδύνους και το καθεξής. Βεβαίως κάποιες δράσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως δεν μπορεί να τις αποδεχτεί μιλώ για την υπογραφή από τους επιτρόπους των διαφόρων ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτας. Δηλαδή, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μάνατζερ και των γενικών διευθυντών είναι συμπληρωματικές με αυτές των επιτρόπων. Δεν είναι ταυτόσιμες. Βεβαίως έχουμε σωστή συνεργασία ώστε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ενήμερη στο επαρκές πολιτικό επίπεδο για, για τα τεκτενόμενα στο επίπεδο το διαχειριστικό, το επίπεδο της διοίκησης και ως σώμα επιτρόπων ε, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή και το πράττουμε άλλωστε να αναλάβουμε πλήρως τις πολιτικές ευθύνες που μας αναλογούν. Τρίτη δράση προτεραιότητας δική σας. Συμφωνούμε ότι η προχρηματοδότηση πρέπει να την χάνει περισσότερο αυστηρής παρακολούθησης. Με τις αλλαγές που έχουμε κάνει στον χρηματοδοτικό κανονισμό θα έχουμε καλύτερη παρακολούθηση των ε, πληρωμών προχρηματοδότησης. Ως προς την τέταρτη δράση προτεραιότητας για ένα αποτελεσματικό μηχανισμό κυρώσεων στη, στον τομέα της πολιτικής συνοχής, θέλω να επαναλάβω τη στεναρή μας δέσμευση να επιτηρούμε εκ του σύνεγγυς τα προγράμματα υλοποίησης όλων αυτών των πολιτικών και να ε, κηρύσουμε αναστολή και πάυση πληρωμών εκεί όπου ε, υπάρχει το πρόβλημα. Ως προς την επόμενη ε, γενιά των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση για τις διορθώσεις βλέπουμε ότι οι θέσεις απομακρύνονται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο από αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Και θέλω να επαναλάβω ε, την έκκλησή μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την πρόταση. Να την στηρίξουν οι πιο βασικές σας επιτροπές, οι οποίες άλλωστε ε, διαδραματίζουν και το ρόλο του συνομοθέτη βάσει της υφιστάμενης νομικής βάσης οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και οι δικές μας εκθέσεις του δικού μας εσωτερικού ελέγχου δείχνουν ότι χωρίς στεναρή δέσμευση από άλλους οικονομικούς φορείς, δηλαδή χωρίς τη δέσμευση των ε, αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, είναι αδύνατο να γίνει σεβαστή η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επομένως τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει μόνο να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και να μοιράζονται τις ευθύνες με την Επιτροπή για σωστή, την ορθή διαχείριση περίπου του 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, αργότερα μέσα σε αυτό το μήνα θα εγκριθεί ο τροποποιημένος κανονισμός, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές για το ρόλο, για τις ευθύνε των διαφόρων φορέων, περιλαμβάνει κυρώσεις έναντι των εθνικών αρχών, οι οποίες δεν καταφέρουν να κάνουν όρθη διαχείριση του προπολογισμού και περιλαμβάνει και σημαντικά μέτρα απλούστευσης περιμένω και πιστεύω ότι όλες αυτές οι δράσεις θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκτέλεσης του προπολογισμού από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Βλέπετε ότι πάρα πολλά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη τα έχουμε ενσωματώσει, ήδη τα έχουμε εφαρμόσει ή έχουμε προχωρήσει στην επεξεργασία τους και στην υλοποίησή τους. Αυτό είναι επιτυχία για τη δική σας Επιτροπή, αλλά δείχνει και τη στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης για το μέλλον των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλο αυτό το εγχείρημα παρακολούθησης δείχνει ότι δρούμε ακολουθώντας τις συστάσεις σας. Και μάλιστα και αυτές που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και ελπίζω αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της δικής μας δουλειάς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικο... Επικοδομητικός διάλογος. Αυτή ήταν η στάση μας και θα είναι η στάση μας στο πλαίσιο της ακρόασης για τη διαδικασία της επόμενης απαλλαγής η οποία θα ξεκινήσει ως ο νουπο. Προσωπικώς παραμένω στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τη συνθετική έκθεση για τη διαχείριση των επιτευγμάτων το 2011 και για την, ε, ε να σας παρουσιάσω και την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Τώρα, για τα επιτεύγματα της διαχείρισης, Management Achievements είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη λογοδοσία και με το εργαλείο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη διαχείρισης των πόρων και ε, επίτευξη των στόχων. Η ανάληψη ευθύνης είναι μια σημαντική δήλωση από πλευράς του σώματος των επιτρόπων και γι' αυτό η έγκριση αυτής της συγκεφαλαιοτικής έκθεσης ε, αποκτά πλήρη ορατότητα, δημοσιεύεται. Δεν είναι μόνο προς ενημέρωση, αλλά είναι και για συζήτηση και για έγκριση με την αποκαλούμενη προφορική διαδικασία. Η έγκριση της εγκεφαλαιοτικής έκθεσης λαμβάνει χώρα μετά από εκτενή διάλογο μεταξύ Επιτρόπου και Γενικής Διεύθυνσης και κάθε Γενικός Διευθυντής υπογράφει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Για όλους αυτούς τους λόγους η έγκριση της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης δεν είναι καθόλου μια τυπική διαδικασία. Είναι μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας ανάληψης ευθύνης και λογοδεσίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από τις αιτήσει εκθέσεις δραστηριότητας, μέσα από τα σχέδια δράσης, ε, ε, περιλαμβάνουμε τα επιτεύγματα σε αυτή την έκθεση και η σχετική έκθεση για το 2011 παρουσιάζει τα επιτεύγματά μας αλλά και τα αδύναμά μας σημεία. Μιλώ για τις 27 επιφυλάξεις που έχουν κατατεθεί για φέτος από τους γενικούς διευθυντές για διάφορα ζητήματα που άπτονται όλων των πολιτικών και που εκπορεύονται από τις, αιτήσεις, από τις εκθέσεις δραστηριότητας. Περιλαμβάνει η έκθεση αυτή τους τομείς πολιτικής αλλά και τις δράσεις για να ανταποκριθούμε στα αδύναμα σημεία που έχουν εντοπιστεί. Αυτή η έκθεση δραστηριότητας είναι πολύ σημαντική πληροφορία και για την αρχή που δίνει την απαλλαγή αλλά και για το ελεκτικό συνέδριο. Η βασικές οδηγίες για τις εκθέσεις δραστηριότητας για το 2011 έχουν τελειοποιηθεί ώστε να υπάρξει περισσότερη ποιότητα και ώστε να είναι πιο εύληπτες και ευανάγνωστες οι εκθέσεις αυτές. Ταυτοχρόνως έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να εναρμονιστούν οι εκθέσεις για τον υπολογισμό του Residual Error Rate ή για τη χρήση ε, των διαφόρων κριτηρίων που έχουν να κάνουν και με την αποκοινού ε, διαχείριση ή την επιμερισμένη διαχείριση. και πάντοτε έχουμε ακολουθήσει τις αρχές της χρηστής ε, δημοσιονομικής διαχείρισης. Έχει γίνει αναφορά και λογοδεσία για τις διαδικασίες ελέγχου για την νομιμότητα και για το τιμή ύπαρξη παρατυπιών στις ε, συναλλαγές αυτές. Βέβαια, οι επιφυλάξεις ε, αυξήθηκαν από πλευράς ποσότητας, ούτως ώστε να ε, πλησιάσουν περισσότερο στα ευρήματα του ελεκτικού συνεδρίου. Συνήθως όμως ε, οι επιφυλάξεις έχουν να κάνουν με τους περίπλοκους κανόνες επιλεξιμότητας ε, για τους δικαιούχους και από τη μη ορθή εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει περισσότερη απλούστευση για το μέλλον και μάλιστα με πολύ φιλόδοξο τρόπο. Η συγκεφαλωτική αυτή έκθεση ρίχνει φως στις πρωτοβουλίες μας και να σας ευφυστήσω την προσοχή σε κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Καταρχάς, ε, περιμένουμε τα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ε, στον ερευνητικό τομέα από το δείγμα, το κοινό δείγμα, το οποίο εισηχθεί σε ολόκληρη την ερευνητική οικογένεια. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, διαίρεση, την ταξινόμηση του οικονομικών καταλόγων, αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Τρίτον, οι εκθέσει των διαρθρωτικών ταμείων προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ε, ε, οικονομικές διορθώσεις ε, και τις αναβολές. τέταρτων στις αιτήσεις εκθέσεις αποδείται μεγαλύτερη σημασία στο πώς ακριβώς οι πολιτικές έχουν προσφέρει ε, προστιθέμενη αξία ε, στην κοινωνία γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, η προετοιμασία των τομεακών προτάσεων για την περίοδο μετά το 2013 είναι καθοριστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω το περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τα σχέση αιτιετούς τους ελέγχους και την αναλογικότητα του κινδύνου. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η συγκυβερνητική αυτή έκθεση έχει βελτιωθεί περαιτέρω και με την βοήθεια των δικών σα των προτάσεων και ετοιμάτων. Πιστεύω ο τρόπο με τον οποίο οργανωμένη σήμερα η έκθεση και οι πληροφορίε που προσφέρει στου ε, άμεσα εμπλεκόμενου ε, σε διάφορου τομεί ε, εκφράστηκαν εδώ επανειλημμένα. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μου χαρά περιμένω να ακούσω από εσά πώς ακριβώς ε, αξιολογείτε εσείς αυτή τη διαδικασία λογοδοσίας και είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω προτάσεις για βελτίωση προς όφελος ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Αρχής Απαλλαγής. Θα αναφερθώ τώρα λιγάκι στην ετήσια έκθεση ιστορικών ελέγχων που έλαβε χώρα το 2011 και που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18, 28 Σεπτεμβρίου ο εσωτερικός ε, ελεγκτής ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 2011 και αναφέρεται στην κατάσταση οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής. Παρουσιάστηκε η έκθεση ε, για να στηρίξει την συγκεφαλωτική έκθεση οι έλεγχοι προτεραιότητας έλαβαν χώρα για να εντοπιστούν κίνδυνοι σφαλμάτων στις χρηματοψηφιακές συνδιαλλαγές, συναλλαγές και διαπιστώθηκε ότι ε, η εφαρμογή και η εκτέλεση ήταν σωστή. Για αυτή τη χρονική περίοδο ο Γενικός Ελεγκτής δεν αναφέρει ε, κάποιες επιφυλάξεις. Το ποσοστό αποδοχής ε, από τις υπηρεσίες ελέγχου των σημαντικών συστάσεων που εκδόθηκαν εξακολουθεί να είναι κοντά στο 100% και Όσον αφορά ε, την ε, ετήσια έκθεση των ε, άμεσα ενδιαφερόμενων, διαπιστώθηκε ότι οι συστάσεις που εκδόθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή οδήγησαν σε καλύτερο έλεγχο και στην Επιτροπή και στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Βέβαια, η Κομισιόν πιστεύει ότι υπολείπεται ακόμα περιτόριο βελτιώσεων σε επίπεδο εκτέλεσης από τις αρχές ελέγχου και με βάση τις συστάσεις που έχουν κατατεθεί. Θα αναφερθώ στα βασικά θέματα που αναφέρει ο εσωτερικό ελεγκτή και θέλω να σα εξηγήσω τι δράσει που ανελήφθησαν για να ε, ληφθούν υπόψη οι συστάσεις η υπηρεσία ιστορικού ελέγχου ε, όσον αφορά τους ε, ελέγχους απόδοσης, τα αποτελέσματα ήταν θετικά, αλλά επισήμανε ότι είναι απαραίτητο οι δραστηριότητες των γενικών διευθύνσεων να είναι αντικείμενο μέτρησης απόδοσης. Επίσης αυτό ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο κατά την οποία τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου είναι όρημα αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους άρα δηλαδή με αυξημένη αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τους διάφορους τομείς πολιτικής, ο εσωτερικός αλλαγκτής υπογραμμίζει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή στρατηγική στον τομέα της έρευνας και συστήνει ουσιαστικό έλεγχο και στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά στην έδρα της αλλά και στις ε, ε, αντιπροσωπείς που την εκπροσωπούν. Και όσον αφορά τις ε, στρατηγικές ελέγχου των διαθετικών ταμείων, αυτές είναι σε σωστό δρόμο. Όσον αφορά τώρα την πληροφορική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια νέα δομή, έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για να εξορθολογήσει τα συστήματά της πληροφορικής και να τα εντάξει καλύτερα σε ένα πλαίσιο. Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δουλειά που έκανε ο εσωτερικός ελεγκτής κατά το 2001 δικά... Ε, είναι συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές για εσωτερικούς ελέγχους. Και πέρα από το να υπάρχει ε, αυτή η συμβατότητα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εσωτερικός ελεγκτής συνέβαλε σημαντικά έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου διαχείρισης της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή καταλήγει στο ότι οι υπηρεσίες της ε, προσέφεραν ικανοποιητικά προγράμματα δράσης παρά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν και μέσα από την Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει τον σωστό έλεγχο της αποτελεσματικής και έγκαιρης εφαρμογής. Φίλιπ ο νέος επικεφαλής της Επιτροπής εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής, είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσετε ίσως σε περισσότερα θέματα που σας απασχολούν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mr. Commissioner, Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά Επίτροπα, αγαπητά μέλη, κύριε Πρόεδρε. Άρχισε δυστυχώς η πτήση μου και δεν κατάφερα να έρθω εγκαίρως για να ακούσω όλους σας. Θα ήθελα όμως να αρχίσω τώρα τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον ε, κύριο Φίλιπ Ταβέρν. Εμπιστευτικές πηγές μου είπαν ότι σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας κύριε Ταβέρν και γι' αυτό το λόγο σας απευθύνομαι στα γαλλικά για να σας πω χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά τον Επίτροπο και εμείς χρειαζόμαστε τις ιδιότητε που βρίσκονται στη συνθήκη τη Λισαβόνας για το έργο της επιτροπή μα, ελέγχου του προπολογισμού. έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογούμενων με αποδοτικό και συνετό τρόπο. Οι πολίτες, ειδικά τώρα σε περίοδο κρίσης, κοιτάζουν πάρα πολύ προσεκτικά ε, το έργο μας, διότι τα χρήματα, τα κονδύλια δεν είναι πλέον αρκετά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα η Επιτροπή αυτή, πιστεύω ότι έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό έργο Υπήρξαν λοιπόν ε, διαδικασίες απαλλαγής και εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Σούλτς, ε, επισήμανε ότι στις αποφάσεις απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιοι όροι που αναφέρουμε, οι όροι αυτοί οδηγούν σε περαιτέρω ε, αύξηση της γραφειοκρατίας. Εμείς καλέσαμε τον πρώτο κ. Σούλτς να διευκρινίσει λιγάκι το θέμα αυτό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για όλες τις προτάσεις βελτίωσης και στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την, με, με τους επιτρόπους. Δυστυχώς εσείς κύριε Σεμέτα δεν ήσασταν παρόν, αλλά ε, οι συνάδελφοί σας και ο κύριος Μπαρόζο ανέλαβαν αυτή την εργασία. Εγώ λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού ε, επισήμανα ότι είμαστε πρόθυμοι να ε, καταθέσουμε προτάσεις που θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία και το κόστος της γραφειοκρατίας τέτοιου είδου προτάσεις τις δεχόμεθα ευχαρίστως. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας απευθύνω αυτές τις προτάσεις προς εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη. Κύριε συνάδελφε Γκάιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά Επίτροπε Σέμετα, αγαπητοί συνάδελφοι, η Αρχίζει η απαλλαγή με, τις, ε, με την συζήτηση επί των ε, γράφων. Είμαστε, κοιτάζουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Και είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και επίσημα και ανεπίσημα με τους συναδέλφους και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκεφαλαιοτική έκθεση είναι ότι οι γενικές, ε, στις γενικές διευθύνσεις διαπιστώθηκε Διαπιστώθηκαν πολύ θετικά αποτελέσματα από το ελεκτικό συνέδριο Και αυτό φυσικά μας χαροποιεί πάρα πολύ. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι η Επιτροπή αντέδρασε πάρα πολύ θετικά στις προτάσεις μας για τις απαλλαγές από το προηγούμενο έτος. Και η Επιτροπή αυτή αλλά και ο εισηγητής ασχολήθηκαν με αυτές τις προτεραιότητες και μεγάλη σημασία είχαν, είχε η εφαρμογή αυτών των προτεραιοτήτων και αυτό αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και φέτος μπορώ να πω ότι από αυτά που βλέπω τα νέα είναι θετικά. Δεν έχει αλλάξει τουλάχιστον δραματικά η κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Να τονίσω βέβαια εκ νέου την επιθυμία του Κοινοβουλίου να διαπιστωθεί μία, τάση, μία μειωτική τάση αυτό δεν το είδαμε τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται δεν θα το δούμε ούτε στη φετινή έκθεση. Πιστεύω πως από αυτά που διαβάζουμε από τη συγκεφαλαιοτική έκθεση της Επιτροπής μπορούμε να καταρτήσουμε μια ημερήσια διάταξη για το έργο της δικής μας Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Υπάρχουν κάποια σημεία, για παράδειγμα το, τα υψηλά ποσοστά σφάλματος στην πολιτική συνοχής, που είναι σημαντικά και πρέπει να εξεταστούν και από εμάς. Και πιστεύω ότι ειδικά ε, στο θέμα των ε, ποσοστών σφάλματων πρέπει να, είναι, πρέπει να ασχοληθούμε πολύ. Η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο ήλεγξε την διαδικασία ελέγχου και τα μέσα που, έχουμε, που είχαμε στην διάθεσή μας Αλλά μειώθηκαν ε, όμως τα κονδύλια της ε, πολιτικής συνοχής, από ό,τι βλέπω. Μετά από συζητήσεις με τους συναδέλφους, βλέπω ότι υπάρχει αποφασιστικότητα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό φέτος και σίγουρα είναι κάτι που θα πράξουμε. Και θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε όσο το δυνατόν διεξοδικότερα γίνεται. Τώρα όσον αφορά το σύστημα διοικητικού ελέγχου στα κράτη-μέλη που έχει λειτουργικά προβλήματα. Αυτό διαπιστώθηκε σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη μετά από έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγκιο. 18 λοιπόν από τα 27 κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτό τον τομέα και για μένα αυτό είναι φυσικά κάτι άσχημο. Φυσικά δεν αποκλείονται από αυτά τα κράτη ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε οι κατοχώρε, ούτε η Γερμανία. Και πραγματικά αυτό οδηγεί στο ερώτημα τι, τι κάνουμε λάθος και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, σε ποιου τομεί, στον τομέα της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής, για παράδειγμα. Και οφείλουμε να ασκήσουμε κριτική στα ελληπή συστήματα ελέγχου. Φυσικά είναι μέχρι ενός σημείου έργο των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών να διεξάγουν τους ελέγχους, όμως κάποια από αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι σε θέση να, τους, να διεξάγουν τους ελέγχους αυτούς όπως θα έπρεπε. Στην έκθεση απαλλαγής, ε, λοιπόν, στη δική μου έκθεση απαλλαγής αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά ο κίνδυνος αυξήθηκε στον τομέα αυτόν και αυτό πρέπει να μας ε, ανησυχήσει. Γνωρίζουμε από τις εργασίες μας ε, ποια, ποιοι τομείς πάσχουν, σε ποιους τομείς πρέπει να πασχίσουμε για βελτιώσεις, σε ποιους τομείς πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο ε, κεντρικά, και πώς, ε, να, πώς, μπορούμε να, πώς θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Και θα ήθελα να ζητήσω από τους αρμόδιους συναδέλφους και από τα άλλα να διεξάγουμε μία διεξοδική και επικοδομητική συζήτηση για αυτό το θέμα. Γιατί οι δημόσιες προμήθειες είναι τώρα κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο με εξαιρετικά πολύ γραφειοκρατία. Δεν, είναι όμως, δεν έχουμε όμως μόνο αυτά τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα της συνοχής, το πρόβλημα της εξωτερικής βοήθειας, του, ελέγχου, του συστήματος ελέγχου διαχείρισης. Υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι δεν λειτουργούν όπως θα θέλαμε. Και αυτό μας επαναφέρει στο θέμα της άμεσης διαχείρισης, διότι τα ποσοστά σφάλματος στα προγράμματα πλαίσιο κινούνται προς μία όχι τόσο θετική κατεύθυνση και αυτό οφείλουμε να το προσέξουμε. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την έκθεση εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, η οποία άρχισε με τους ελέγχους απόδοσης και αυτό το θεωρώ πολύ σωστό. Η έκθεση αυτή όμως συμπεριλάμβανε και μια και έναν έλεγχο για την διεξαγωγή των ε, δημόσιων προμηθειών. Τα αποτελέσματα του εσωτερικού αυτού ελέγχου για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι οι δημόσιες προμήθειες είναι ένα επίμαχο ζήτημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ποσοστά σφαλμάτων και κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητή, κύριε Γκάιερ. Η συνάδελφος κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σε πολύ σωστό χρονικό σημείο παίρνω το λόγο. Άκουσα τον συνάδελφο από την Επιτροπή ΙΝΚΟ, ο οποίος ασχολείται εδώ και 8 χρόνια εντατικά με το θέμα των δημόσιων προμηθειών. και εκτός από αρκετές περιπτώσεις κρατών μελών όπου οι κανόνες δεν είναι μόνο περίπλοκοι, αλλά παρατηρούνται και εγκληματικέ ενέργειες όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες κατέληξαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις SD που κατέληξαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή σε διαιτησία. Η διαδικασία απλοποίησης δεν θα διαρκέσει μόνο δύο χρόνια, όπως ευχόμαστε, αλλά έξι χρόνια. Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να μας δώσει τροφή για σκέψη. Τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις. Μία βασικά ερώτηση στον κύριο Πίτροπο. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα όσον αφορά τα διαρθρωτικά ε, ταμεία να σας δώσω το εξής. Μας είπατε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία κατευθύνονται σε σωστό δρόμο. Εγώ αυτή τη δήλωση τη βρήκα κάπως λίγη, ελλειπή για την Επιτροπή αυτή. Ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού μας. Και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε για τα τελευταία 1-2-5 χρόνια μας καταδεικνύουν μία ανάγκη για μεταρρύθμιση των διαθροτικών ταμείων. Τι έχει γίνει λάθος λοιπόν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκρέσλε τώρα. Ναι, Κύριε Πρόεδρε, να παραδεχτώ ότι δεν επεξεργάστηκα εντατικά τα έγγραφα. Με απασχόλησε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου δυστυχώς τον τελευταίο καιρό και δεν κατάφερα να τα μελετήσω με εξαιρετικές λεπτομέρειες. Ένα ερώτημα έχω, ιδιαίτερα εν ώψη των δραματικών εξελίξεων στις χώρες της Ευρωζώνης. Η πολιτική μας στόχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Και ήταν και τον, ε, το απερχόμενο έτος. Τι γίνεται φέτος. Επίσης, η αιτήσια, η έκθεση πεπραγμένων, στην έκθεση αυτή βλέπω ότι έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος κινηθήκαμε και αυτό να το αναγνωρίσω και να το συγχαρώ, όμως πραγματικά θα πρέπει να, πραγματικά να ρωτιέμαι πώς θα γίνει η δημοσιονομική εξυγίανση των κρατών μελών σε συνδυασμό με, τον, ε, με την ευρωπαϊκή εξυγίανση των δημοσιονομικών. Εάν δεν καταφέρουμε να εξηγιάνουμε τα δημοσιονομικά με ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε το πρόβλημα θα γιγαντωθεί και δεν θα έχουν πρόβλημα μόνο με μονομένα κράτη-μέλη, αλλά όλη η Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την απαλλαγή, τι κάνουμε με τα χρήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς τα χρησιμοποιούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επιδεινώσουμε επίσης την κατάσταση και έπειτα όσον αφορά το σύστημα Γκαλιλαίο. Πώς βλέπετε το μέλλον του συστήματος Γαλιλαίου με τα προβλήματα που έχουν προκύψει και τι κάνετε για να βελτιώσετε και να λυπηλήσετε τα προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα οποία είπαν οι τρεις ε, συνάδελφοι. Υπάρχει λοιπόν το θέμα ε, του ελέγχου και των ε, χρηματοδοτικών ε, διορθώσεων. Αυτό για μας ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν θέμα ουσίας και πραγματικά εκπλαγήκαμε για το ότι το Συμβούλιο το θέμα το αντιμετώπισε διαφορετικά. Εκπλαγήκαμε για το ότι ήταν δύσκολο να επιτευχθεί η συμφωνία και το ότι μάλιστα υπήρξαν χώρες ε, οι οποίες ε, τώρα στις ε, διαβουλεύσεις για τον προεπολισμό τάσσονται υπέρ του περίφημου better spending. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο κύριος Ρομπέ με τον οποίο συζήτησα μίλησαν για αυτό το θέμα, για τον έλεγχο του προπολογισμού, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πώς μπορεί αυτό να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. Κατατέθηκαν λοιπόν προτάσεις, ε, όπως είπε και η κυρία ε, Γκρέσλε, για ένα ειδικό προπολογισμό. Αυτό όμω ε, δεν είναι προ όφελο ούτε του δικού μας του Κοινοβουλίου, ούτε προ όφελο του φορολογούμενου. Εφόσον υπάρχει κοινοβούλιο, μπορεί να λάβει και αυτό το καθήκον. Ίσως λοιπόν, κύριε Επίτροπε, μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού του θέματος, να μας πείτε τη δική σας την άποψη ή ίσως ε, στο Σώμα των Επιτρόπων να έχει ε, διαμορφωθεί κάποια επικρατούσα άποψη. Και αν θέλετε βέβαια προφανώς μπορείτε να τοποθετηθείτε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις που ετέθησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ε, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ευρύτερο θέμα σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στην συνεισφορά του προϋπολογισμού στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει κάποια παρεξήγηση σχετικά με το νόημα του κοινοτικού προπολισμού. Το νόημα ε, του κοινοτικού προπολισμού είναι ε, να υπάρξουν επενδύσεις. Είναι επένδυση στην ανάπτυξη και στις ε, θέσεις απασχόλησης. Ο κύριος Χάν, όταν θα έρθει εδώ, θα σας εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που σας είπα. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, ο κοινοτικός προπολογισμό συμβάλλει μέχρι και 75 ή 90% του συνόλου των επενδύσεων. Άρα δηλαδή χωρίς τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τον ενωσιακό, θέλετε, ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επενδύσεις ε, στην υποδομή, ε, σε προγράμματα ανάπτυξης. Ξέρω, ας πούμε από το δικό μου, από τη δική μου την πατρίδα, το 80% των επενδύσεων χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατανοούμε τα αιτήματα μερικών κρατών στην όλη συζήτηση που γίνεται για το επόμενο πολίτες ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που λένε ότι να υπάρξει μείωση των προτάσεων της Κομισιόν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι απολύτως γανθασμένη στάση και μάλιστα αυτή είναι αντίθετη με τον ευρύτερο στόχο μας που είναι να προάγουμε την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης στα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή σχετικά με την μεγαλύτερη, περισσότερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο μάλλον στην Ευρωζώνη, για να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα αυτής. Βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι μας ότι διεξάγονται συζητήσεις, τουλάχιστον στον δημόσιο τομέα, για να διαπιστωθεί κατά πόσον ε, η, Ευρωπα... η Ευρωζώνη θα μπορούσε να έχει το δικό της τον προπολογισμό. Γίνεται αυτή η κουβέντα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρί ε, για να συζητήσουμε λεπτομέρειες αυτής της ιδέας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο προεδρεύων του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, της Ευρωζώνης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλοι αυτοί οι πρόεδροι, μα πέντε πρόεδροι, αυτή τη στιγμή συζητάνε αυτό το θέμα και όταν ε, θα καταθέσουν τις απόψεις τους Ελπίζω αυτό να γίνει ε, κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τότε λοιπόν ε, θα έχουμε και εμείς κάποια βάση για να γίνει συζήτηση επί του θέματος πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ερωτήσεις του κυρίου Γκάια. Σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και στους ελέγχους που αφορούν στις κρατικές, στις δημόσιες προμήθειες. Το αποτέλεσμα αυτών των, αυτού του ελέγχου ε, κατατέθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου Πρόοδου ελέγχου και έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της ε, υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Αυτές λοιπόν οι συστάσεις σε μεγάλο βαθμό θα συμβάλλουν στο να διαμορφωθούν οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με νέους κανονισμούς για τις κρατικές προμήθειες. Α, από την άλλη, η Γενική Διεύθυνση Αγορά δεσμεύτηκε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην εφαρμογή κανόνων για τις κρατικές προμήθειες και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά στην διαδικασία απαλλαγής ε, για φέτος, είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε τι θα περιλαμβάνει η έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, στην Επιτροπή βλέπουμε ότι, είναι, ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα λάθη στις ε, κρατικές προμήθειες και αυτά δεν οφείλονται στην κοινοτική αλλά στις εθνικές νομοθεσίες που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη επιβάλλουν στις εθνικές νομοθεσίες εφαρμοστικούς κανόνες οι οποίοι ε, δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται σεβαστοί. Όσον αφορά τώρα ε, τους ελέγχους απόδοσης, κύριε Γκάια αναφέρατε ότι αυτό είναι μια ε, πολύ ευχάριστη εξέλιξη και μάλιστα η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποδίδει όλο και μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο απόδοσης. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα ε, θα οργανωθεί ένα συνέδριο ε, το οποίο θα ασχοληθεί ακριβώς με θέματα ελέγχου απόδοσης. Και αυτό θα λάβει υπόψη του την ανάγκη να υπάρξουν αποτελέσματα όσον αφορά στους ε, ελέγχους. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Βάιλα σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι ίσως σήμερα είναι πολύ νωρίς για να αναφέρει κανείς τα αποτελέσματα ε, του 2011 τα απορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Απλά θέλω να πω ότι η δική μας δράση αφορά ε, στην αυστηρή ε, φαρμογή, στην αναστολή καταβολών, στην διακοπή καταβολών, πληρωμών και αυτά όλα έχουν ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, τις δραστηριότητες μας αυτές ε, και μάλιστα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για πρώτη φορά ε, συμμετείχε στον έλεγχο εθνικών αρχών ελέγχου στα κράτη-μέλη. Διότι βεβαίως ένα από τα προβλήματα που υφίστανται είναι ότι οι εθνικοί οργανισμοί ελέγχου δεν είναι απόλυτα σε θέση να διεξάγουν ελέγχους υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να εξευρεθούν τρόποι να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητά τους. Ε, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι Υπάρχει το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο ελέγχου. Αυτά βέβαια τα επίπεδα προφανώς είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, κατόπιν τούτου ε, και εμείς οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η επόδοσή τους. Προσβλέπουμε βέβαια στην, ε, στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε νέα προγράμματα όπου προτείνουμε ε, αυστηρά μέτρα σχετικά με καθαρές ε, διορθώσεις. Αυτό είναι ένα τελείως νέο φαινόμενο, αλλά είναι πολύ σημαντικό η πρόταση αυτή της Κομισιόν για καθαρές διορθώσεις να στηριχθεί και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω βέβαια ότι πέρυσι η Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών ε, υποστήριξε στεναρά αυτήν την πρόταση και στις άλλες επιτροπές όμως δυστυχώς καταβάλλονται προσπάθειες να αποδυναμωθεί αυτή η έκθεση. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε μία συνέπεια στη συμπεριφορά όσον αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Και τέλος όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε σχετικά με το πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πέρυσι διεξήγε διάφορους ελέγχους σχετικά με το πρόγραμμα αυτό και συζητήσαμε τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων στην Επιτροπή ε, Πρόοδου Ελέγχων. Και το πρώτο που κάναμε ήταν να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη διαχείριση αυτού του προγράμματος. Τώρα υπάρχει ένας αναπληρωτής γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει επιληφθεί του προγράμματος και όλες οι συστάσεις ε, που ε, κατατέθηκαν από την Υπηρεσία Ιστορικού Ελέγχου έγιναν αποδεκτές από αυτή τη Γενική Διεύθυνση που σας προανέφερα. Γιατί στόχος είναι η ενίσχυση της διαχείρισης, βεβαίως και Υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, όμως ε, αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στον, στην αποτελεσματική διαχείριση. Και αν γίνει αυτό, αναμφίβολα θα αμβληνθούν οι κίνδυνοι που απειλούν το πρόγραμμα ε, Γαλιλαίος. Νομίζω ότι απάντησα σε όσες ερωτήσεις μου τέτοια μέχρι τώρα. Yes, thank you very much. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Επομένως, Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Γκάγερ που είναι ο εισηγητής θέλει όμως ε, να ξανασχολιάσει. Όχι. Μάλιστα, τότε μπορώ να ολοκληρώσω τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ανυπομονούμε για τις ε, επερχόμενες συζητήσεις για την έκθεση. Ξανά κύριε Ταβέρν, χρόνια πολλά για σήμερα. Στρογγυλό αριθμό κλείνεται. Και επίτροπε έμετα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω. Περνάμε σε, σε θέματα όχι και τόσο εύκολα την καταπολέμηση της απάτης. Θα ήθελα να σας δώσω τώρα το λόγο για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να, στρα... να σχολιάσω το δεύτερο, σήμερα... το δεύτερο ζήτημα για το οποίο ήρθα να σας μιλήσω οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης η οποία έχει αντίκτυπο στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκάιερ την επόμενη εβδομάδα θα διοργανώσει μια ακρόαση ε, για το θέμα αυτό, την οποία και θα παραστώ, αφού με κάλεσε και τον ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ωστόσο, επειδή θα πρέπει εκείνη τη μέρα να ταξιδέψω στην Ινδία, ε, θα ε, έρθει προς αντικατάστασή μου ο κύριος Κέσλερ, ο Γενικός Διευθυντής. Το θέμα λοιπόν της ε, ε, καταπολέμησης της απάτης είναι ένα θέμα το οποίο με αγγίζει πραγματικά και σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω τις πρωτοβουλίες που έχω ήδη ξεκινήσει στον τομέα αυτό, αλλά και τις επικείμενες πρωτοβουλίες που προτίθεμαι να αναλάβω. Πρώτο σχέδιο, πρώτο πρόγραμμα το έχουμε ήδη αναφέρει στην Επιτροπή σας σήμερα. Χαίρομαι διότι εγκρίνατε τη συμβαστική λύση που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές για την τροποποίηση, για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού της Όλαφ. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτή η συμφωνία και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε διότι πράγματι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να κλείσει το θέμα. Η μεταρρύθμιση της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της απάτης είναι μια μεταρρύθμιση που συζητούμε τα τελευταία έξι χρόνια και παραπάνω. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης. Ο νέος κανονισμός θα διευκρινίζει τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και θα επιτρέψει πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ήδη ανα, αναφέρθηκα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ψηφοφορία του κανονισμού της Όλαφ. Δεν θα τα επαναλάβω βεβαίως. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της Όλαφ ήταν στην ημερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι επόμενες πρωτοβουλίες στις οποίες θέλω να αναφερθώ είναι πολύ πιο πρόσφατες ή είναι και επικείμενες. Τον Ιούλιο του 2011 καταθέσαμε μια πρόταση οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του ποινικού δικαίου. Είναι μια πρόταση από κοινού που έχουμε κάνει εγώ και η Επίτροπος κυρία Ρέντιν για να αναρμονιστεί και να ενισχυθεί το ποινικό δίκαιο στα κράτη-μέλη ως προς τα δικήματα που διαπράττονται ενάντια και καταφέροντας πλήγμα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, Γιατί είναι διαφορετικά τα επίπεδα προστασίας στα κράτη-μέλη ως προς το θέμα αυτό. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα παράδειγμα να καταλάβετε καλύτερα. Από το 2000, 281 από τις 647 υποθέσεις, 281 από τις 687 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν από την Όλαφ στις εθνικές υπηρεσίες τελικά έκλεισαν ως ε, θέμα. Δεν, ε, δεν βγήκε κανένα πόρισμα, δεν έγινε καμία παρακολούθηση και δεν επιτεύχθηκε και τίποτα. Από το 14 μέχρι το 80% λοιπόν κυμαίνεται αυτό το ποσοστό των υποθέσεων που μπαίνουν στο αρχείο και μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς να βγάλετε το μεσοόρο. Η οδηγία που προτείναμε τον Ιούλιο λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, καλύτερος ορισμός των αδικημάτων που καταφέρνουν πλήγμα στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι με τον ίδιο τρόπο γίνεται αντιληπτή η ποινικό κολάσιμη συμπεριφορά σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ελάχιστες κυρώσεις για τα εν λόγω ώστε να έχουμε ισοδύναμη, αναλογική αλλά και επαρκή επιβολή κυρώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, επέκταση των περιορισμών, των καταστατικών περιορισμών, ώστε οι ερευνητές, οι εισαγγελείς, ε, οι ανακριτές έχουν αρκετό χρόνο να διενεργήσουν διασυνοριακούς ελέγχους και έρευνες πιο ενδελεχώς και πιο λεπτομερώς. Την πρόταση αυτή την έχουμε διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και βασίζομαι στη στήριξή σας για τη γρήγορη έγκριση και υιοθέτησή της. Και μάλιστα αυτή η γρήγορη έγκριση είναι πολύ πιο σημαντική διότι εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του πώς θα επανασχεδιάσουμε ε, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Τον Ιούνιο ε, προτείνουμε να, ε, σκοπεύουν να προτείνουμε ε, τη δημιουργία του EPPO, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό γραφείο, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία εισαγγελικών αρχών, Public Prosecutor Office, European Public Prosecutor Office. Θα έχουμε και πρόταση μεταρρύθμισης του Eurojust και έτσι θα ολοκληρώσουμε όλο αυτό το νομοθετικό πακέτο θα γνωρίζετε ότι η δυνατότητα σύστασης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Δημοσίου Εισαγγελέα Πολιτικής Αγωγής ε, είναι κάτι που από την Eurojust είναι κάτι που προβλέπεται στη συνθήκη, την τελευταία συνθήκη που έχει υπογραφεί για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχει διδάξει εμπειρία ότι η εθνική εδαφικότητα και η εθνική νομολογία δεν αρκεί ως πλαίσιο για να επιλύσουμε περίπλοκες υποθέσεις οι οποίες εκφύσεως είναι ευρωπαϊκές και ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Έτσι όπως έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, ε, δεν είμαστε σε θέση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος των προκλήσεων που ε, γύρει μπροστά μας το διεθνές και το οργανωμένο έγκλημα και αυτό είναι απαράδεκτο πόσο μάλλον αφού διανύουμε περίοδο οικονομικής ε, και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν να στηρίξουμε την ανάπτυξη, να καταπολεμήσουμε ε, την παραοικονομία και να μην αφήνουμε τον κάθε έναν να ε, τσεπώνει χρήματα και να μας ξεφεύγει. Η Όλαφ λοιπόν μπορεί να διενεργήσει ε, διοικητικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της απάτης. Το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα ε, θα μπορεί να διενεργεί πολύ πιο εκτεταμένες έρευνες και να απαγγέλει ποινικέ ε, κατηγορίες και να ασκεί ποινικέ διώξεις όταν διαπράττονται αδικήματα ενάντια στο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διερευνήσει και να ε, εξηχνιάσει περίπλοκες υποθέσεις απάτης. Και γι' αυτό οι υπηρεσίες μας εξετάζουν διάφορες αναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Από την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2001 μέχρι και σήμερα έχουμε κάνει προπαρασκευαστική έρευνα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο. Η πρόταση της ε, Κομισιόν λοιπόν θα βασίζεται σε αυτή τη δουλειά ε, και σε μια λύση η οποία θα έχει την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλειας. Πέρα από τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εισαγγελικών Αρχών, ε, δημοσίου κατηγόρου αν θέλετε, θα έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε ρυθμίσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή βελτίωση πληροφοριών σε έρευνες οι οποίες είναι πολυτομεακές, έρευνες ε, που απαιτούν τη συνεργασία διοικητικών αρχών, φορολογικών αρχών, αστυνομικών αρχών, τελωνιακών αρχών και δικαστικών αρχών ενδεχομένω. Αυτά είναι πρόκληση αυτός ο συγκερασμός και ο συνδυασμός όλων αυτών των διαφορετικών αρχών. Δεν πρέπει όμως να είμαστε μη αποτελεσματικοί. Πρέπει να έχουμε υψηλές επιδόσεις για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε θα πρέπει και εμείς λοιπόν να γνωρίζουμε σύνορα. Όλα αυτά τα μέσα θα διευκολύνουν τη δουλειά ε, του EPPO, της υπηρεσίας αυτής της οποίας τη σύσταση θα προτείνουμε. Είναι πολύ σημαντικά στο εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Και τελευταία από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε είναι η εξή, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντική, το ίδιο σημαντική αν όχι περισσότερο, ε, ε, για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και αναφέρομαι στην προστασία του ευρώ. Οι συζητήσεις με τους εμπειρογνωμόνες μας μας έχουν δει δείξει ότι δεν θα πρέπει να μας νοιάζει μόνο η οικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, θα πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία των χαρτονομισμάτων και κερμάτων ε, ε βάσει και του ποινικού δικαίου. Δηλαδή όλες οι αρχές, τα κράτη-μέλη, να μπορέσουν να, να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τις ερευνητικές που διατίθενται για άλλα δικήματα του οργανωμένου εγκλήματος και σε αυτή την περίπτωση και για τα του ευρώ θέματα των ε, και νομισμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω τις μη νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Θα θυμάστε ότι το περασμένο καλοκαίρι οι υπηρεσίες μου προέβαλ, πρότειναν το σχέδιο δράσης ανατολικών συνόρων προκειμένου να καταπολεμηθεί το ελαθρομπόριο καπνού και τσιγάρων στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκτοτε αυτό είναι προτεραιότητά μου. Το λαθρεμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και τσιγάρων στοιχίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 10 δις ευρώ το χρόνο, τα οποία χάνονται. Και μάλιστα ε, σε καιρού τόσο ε, σφιχτής δημοσιονομικής διαχείρισης, αυτά είναι ποσά ε, που δεν, μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιτρέπουμε στους εαυτού μα να μην τα εισπράττουμε και να τα χάνουμε. Έχουν δείξει τα τα στοιχεία και οι έρευνες ότι έχει κάπως ειρικνωθεί αυτή η λαθρέα η παραοικονομία, η παράνομη αγορά. Ωστόσο, σε μέγεθος, σε όγκο, σε κύκλο εργασιών εντός εισαγωγικών, αλλά ε, η δραστηριότητα δεχομένω αυξάνεται ο, στις χώρες της Βαλτικής. Η KPMG στην έρευνά της μας έχει δείξει και έχει βρει στα απορίσματά της ότι ε, στις χώρες του Νότου το λαθρεμπόριο από 13% το 2010 έχει πάει στο 19% το 2011, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της KBMG το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και τσιγάρων και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί. Στόχος μας είναι να έχουμε μια ε, στρατηγική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θα περιορίζεται στα ανατολικά, στα ανατολικά σύνορα. Ε, βρισκόμαστε σε πρωταρχικό στάδιο ε, της δουλειάς μας και το πρώτο μισό του 2013 θα υποβάλω αυτές τις προτάσεις και στους υπόλοιπους επιτρόπους. Ε, πρόθεσή μας είναι να εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένουμε τα ε, δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτάσεις, τη δική σας ε, συμβολή. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Όλαφ συνεργάζεται με άλλους φορείς για το μηχανισμό υποβολής αναφορών κατά της διαφθοράς. Είναι κάτι που επινοήθηκε και συστάθηκε το 2011, τον Ιούνιο. Η Συνάδελφο Σεσίλια Μάιλστρομ και η Γενική Διένθεση Αρμόδια για Εσωτερικές και Νομικές Υποθέσεις έχουν ε, ε, τεθεί επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας. Ε, η πρώτη έκθεση θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013 και θα περιλαμβάνει γενικότερα θέματα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο ειδικά θέματα ανά χώρα και εκεί θα έχουμε μια πιο ενδελεχή ανάλυση. Οι συστάσεις δεν θα είναι νομικώς δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη, ωστόσο θα κάνουμε την παρακολούθηση και θα δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους για πάνω σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ανατέθηκε στην Όλαφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βασικό στόχος είναι να καθοριστεί μια μεθοδολογία για να υπολογιστεί το κόστος της διαφθοράς στις κρατικές προμήθειες ή στις δημόσιες αγορές αν θέλετε. Και αυτό το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη ε, του χρόνου. Αξιότιμα μέλη, ελπίζω, νομίζω ότι κατάφερα να παρουσιάσω μια επισκόπηση των πιο σημαντικών υφιστάμενων αλλά και, αλλά και μελλοντικών πρωτοβουλειών ώστε να προστατευθούν ε, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πολλά άλλα πράγματα ε, κάνουμε ε, στις υπηρεσίες μας. Έχουμε και την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, με εσάς τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Αρχίζουμε με τον εισηγητή κύριο Γκάιερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Επίτροπε κυρία Σέμετα, για την παρουσίαση. Πιστεύω πως μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά έχει καταπιαστεί με όλες τις πτυχές του ζητήματος και αυτό το χαιρετίζω. Πράγματι θέσαμε προκαιρού αυτό το ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και το έργο της και εν λοιπόν αυτού και εν των ε, αριθμών που έχουμε στη διάθεσή μας όσον αφορά την απάτη στην Ευρώπη. Και από ό,τι βλέπω είτε είναι λοιπές στο νομικό πλαίσιο είτε λυπή η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αντιμετωπίζουν την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορές από κράτος ε, σε κράτος. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαδικασία, το έργο της Όλεφ έχει συναντήσει προβλήματα. Πιστεύω πως πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε το έργο της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με ανησυχεί όμως σε αυτό το, σε αυτό το ενισχυμένο νομικό πλαίσιο που θέλουμε να καταρτήσουμε. Μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο παρακολύσεως παρεμποδίσεως το, του έργου των κρατών μέλων και πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Τα κράτη-μέλη πραγματικά θα πρέπει να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα το νομικό πλαίσιο δίνοντάς του την πρέπουσα προσοχή. Με ανησυχεί λοιπόν αυτή η εφαρμογή όπως σας είπα και ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνδεσή της με το πολιετές σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακριβώς γιατί υπάρχει απάτη, υπάρχουν ποσοστά ασφάλματος στις ε, μεταφορές, υπάρχουν σφάλματα στον προϋπολογισμό. Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ξεκάθαρο στα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται βελτίωση. Με χαροποιεί πάρα πολύ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολιτική συζήτηση με εμάς. Η ερώτησή μου όμως σε όλους τους συναδέλφους είναι εξής. Τι κάνουμε εάν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να συμπεριφέρονται όπως φοβόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος συνάδελφος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίτροπο για τις πρωτοβουλίες αυτές για το μέλλον. Στηρίζω επίσης να πω και τον συνάδελφο Γκάιερ, ο οποίος εξέφρασε τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του για τις ε, Νομικέ πρωτοβουλίε και για το ότι αυτέ ίσω δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της απάτηση. Εντάξει, βέβαια, αυτό που γίνεται για την καταπολέμηση της ε, εισαγωγή λαθρέων τσιγάνων στα ανατολικά σύνορα είναι καλό. Αλλά σήμερα το 40% των τσιγάρων που καταναλώνονται στην Λιθουανία είναι λαθρέα. Επίσης αναφέρθηκε ότι το παραεμπόριο αυτό μεγαλώνει, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη στη Νότια Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερωτώ με, θα ήταν καλό να ενισχύσουμε το ποινικό υπόλογο και αν ναι, χρειάζεται να αναφέρουμε σαφώς και ρητά ποιες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες στα κράτη-μέλη. Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε τις εκθέσεις στη διάθεσή μας. αλλά θα έχει περάσει ένα μισή χρόνο από το 2011 και οι παρατάσεις αυτές ε, συνεχίζονται και από χρόνο σε χρόνο και διαιωνίζονται και θα υπάρχουν θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη που θα είναι υπεύθυνε για το λαθρεμπόριο και την απάτη θα υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες που θα έχουν εντολή και ευθύνη να επιληφθούν του θέματος και αυτό φυσικά ε, να τονίσω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα καλύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Τεό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, με συγχωρείτε, είχα ένα τηλεφώνημα. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε είναι υψή της σημασίας και χαίρομαι πάρα πολύ που ενημερωθήκαμε από τον κύριο Πίτροπο γι' αυτό. Είναι σαφές ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα για την Επιτροπή μας. Υιοθετήσαμε επίσης και μία, ε, έχουμε όμως και μία έκθεση για το ποινικό δίκαιο και υπάρχουν τμήματα εκεί που αφορούν αυτή την Επιτροπή. Είναι σημαντικό πιστεύω να τονίσουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό και σημαντικό και ότι είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε σε ευρωπαϊκό, σε κοινοτικό επίπεδο και όχι κάθε κράτος μέλος μόνο του. Αυτό παρουσιάζεται και στο επεξηγηματικό σημείωμα. Αυτό που δεν έχω δει όμως είναι μια εκτίμηση αντικτύπου, η οποία να έχει τα νούμερα και να μπορέσει να με πείσει ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εφαρμόσιμο. Το Κοινοβούλιο πραγματικά χρειάζεται πολλές πληροφορίες από αυτού. Αυτός είναι και ο, αυτή είναι και η σωστή οδό. Αυτό προσδίδει προστιθέμενη τη θέμενη αξία. Διότι φυσικά το θέμα του ποινικού δικαίου και των ε, ποινικών κυρώσεων είναι πολύ ευαίσθητο και η πρόταση αυτή θα έχει εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Τότε θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πίτροπο να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με την τελευταία ερώτηση που αφορά την εκτίμηση αντικτύπου. Κάθε πρόταση, κάθε τόσο σημαντική πρόταση, φυσικά και χρειάζεται εκτίμηση αντικτύπου. δρομολογείται αυτό και έχουν γίνει διεξοδικές εκτιμήσεις αντικτύπου οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποινικό δίκαιο. Μπορούμε λοιπόν να σας παρέχουμε αυτές τις εκτιμήσεις αντικτύπου αλλά και τις ε, μελλοντικέ όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελικών Αρχών. Ε, αναμένουμε την εκτίμηση αντικτύπου πάνω σε αυτό, καθώς και για την πρωτοβουλία όσον αφορά την ποινική δικονομία. Κάθε πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία που ανέφερα σήμερα, φυσικά και θα υποστηρικτεί από διεξοδικότατες εκτιμήσεις αντικτύπου και θα τις παρουσιάσουμε εδώ ενώπιόν σας, γιατί συμφωνώ μαζί σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αποφάσεις σας να είναι βασισμένες σε μια διεξοδική ανάλυση, η οποία θα έχει γίνει από εμπειρογνώμονες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που έθεξε ο κύριος Γκάιε για το πόσο εφαρμόσιμη είναι οι κανόνες σε επίπεδο κρατών μελών. Ακούστε. Πιστεύω πως αυτό το πακέτο, αυτό το σύνολο, τη δέσμη μέτρων που προτείνουμε, θα είναι η βάση για το νομικό πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελικών Αρχών, δεν θα είναι οδηγία αλλά κανονισμός. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν ως οδηγία να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή δικονομικούς κανόνες για το ποινικό δίκαιο. Άρα αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα από τα ζητήματα που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και που έχει συμβάλλει και στα νούμερα που σας παρουσίασα. Όταν παρουσιάζονται οι υποθέσεις που αναλαμβάνει η Όλευ στα κράτη-μέλη, αυτά τα κράτη-μέλη δηλαδή, δεν τις αναλαμβάνουν από την αρχή. Γίνεται δηλαδή αυτή η έκθεση, μετά πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Και σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη αρχίζουν από την αρχή έρευνες. Αυτό λοιπόν όπως καταλαβαίνετε είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και το καθιστά λιγότερο αποδοτικό. Και προσπαθούμε με την δικονομία να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις της Όλαφ αποτελούν την αφετηρία των ερευνών εκάστοτε υπόθεση απάτης. Όσον αφορά το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Μπαλτσίτου, θα ήθελα να πω ότι καταρχάς το λαθρεμπόριο τσιγάρων και τα σχετιζόμενα με αυτό ζητήματα δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών αυτό. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουν το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Φυσικά, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αρμοδιό... τις αρμοδιότητες που έχουμε μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω πως θα ήταν θεμελιωδώς λάθος το σκεπτικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λύσει τα προβλήματα παραποίησης που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος. Αυτό δεν γίνεται, δεν θα συμβεί. τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ε, ευθύνε τους για το έργο αυτό. Τώρα όσον αφορά το, τα νούμερα που μας είπατε, το 40% για παράδειγμα των ε, τσιγάρων που καταναλώνονται στην Λιθωνία, αν δεν κάνω λάθος, είναι λαθρέα. Εγώ θα πρότεινα να κοιτάξετε τις ε, νεότερες εκθέσεις, εκθέσεις εκτίμησης για τις παράνομες αγορές, αγορές παραποιημένων προϊόντων. Και στη Λιθουανία από το 40% το ποσοστό λαθρέων μειώθηκε στο 20, 9% κατά 11 ποσοστίες μονάδες δηλαδή. Αυτό είναι στην μελέτη. Φυσικά είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, δεν σημαίνει βέβαια ότι λύσαμε το πρόβλημα. των παραποιημένων προϊόντων στα κράτη-μέλη. Και όπως ανέφερα και στην εισαγωγική μου ομιλία, αυτό το φαινόμενο είναι κάτι καινούριο. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας στα ανατολικά μας σύνορα. Και ακριβώς επειδή ενισχύσαμε τις προσπάθειες αυτές, βλέπουμε ότι η ροή κατευθύνθηκε προς τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγονται από εκεί τα λαθρέα τσιγάρα δηλαδή και τα υπόλοιπα παραποιημένα προϊόντα. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε την ασφάλεια των συνόρων σε όλο το εύρος τους, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, ίσως δεν κατάλαβα κάτι καλά. Αλλά στους κανονισμούς της Όλαφ προβλέπεται η ανάγκη τα κράτη-μέλη να αναθέτουν την αρμοδιότητα στο εκάστοτε συντονιστικό όργανο που θα λειτουργεί σε κάθε κράτος μέλος και θα συνδέεται με την Όλαφ. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θα συντονίζουν την ε, δραστηριότητα της ε, καταπολέμησης της απάτης. Νομίζω πως ε, κάλυψα τις ερωτήσεις και είμαστε στη διάθεσή σας και για περισσότερες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιος άλλος το λόγο. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τουλάχιστον τη στιγμή όχι. Αλλά θα ήθελα όμως ε, να δράξω την ευκαιρία, πριν δώσω και το λόγο και πάλι στον Αλφα Βαλτσίτης, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά τον πρόεδρο της ε, Όλαφ, τον κύριο Κέσλα. Κύριε Κέσλα, είστε πάντα ευπρόσδεκτος και ειδικά στο θέμα αυτό. Ε, αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι τι ρόλο παίζει η Όλαφ και πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και αν υπάρχουν ερωτήσεις και ο κύριος Κέσλε είναι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα όμως καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Labai žingsniai buvo padaryti dėl kontrabandos mažinimo Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατορθώσαμε να περιορίσουμε ε, τις, ε, τον όγκο το, του λατρεμπορίου τσιγάρων, αλλά ε, Υπάρχουν βέβαια τα στοιχεία της Φίλιπ Μόρις. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, η στρατηγική για το μέλλον για την αντιμετώπιση της απάτης και του λαθρεμπορίου. Υπάρχει μια τέτοια στρατηγική, αλλά θέλω να πω ότι στα κράτη-μέλη επικρατεί χάος, γιατί ο ορισμός ε, του λατρεμπορίου δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να προβεί κανεί σε κοινέ ενέργειες. Προφανώς ε, σήμερα δεν ε, ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά κύριε Επίτροπε, δεν θεωρείτε και εσείς ε, ότι θα ήταν σκόπιμο να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ορίσουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να οριστούν και οι αρμοδιότητες. Θα μου δώσετε λοιπόν την ευκαιρία να απαντήσω κι εγώ στη μητρική μου γλώσσα, λέει ο Επίτροπος. Βεβαίως ε, υπάρχει η αρχή της ε, επικουρικότητας. Και δεν μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιβάλλουμε το τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Πάντως, κατά τη δική μου άποψη, αυτά τα οποία εφαρμόζονται μέσα από το πρόγραμμα δράσης για τα ανατολικά σύνορα, αυτά έχουν ήδη αποφέρει αυτά αποτελέσματα. Μπορούμε να δούμε την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους ε, διάφορους οργανισμούς ε, και στα κράτη-μέλη και στα σύνορα και διασύνοριακά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση τώρα πια είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Βεβαίως και θα επιθυμούσαμε να εξαλείψουμε το λαθρεμπόριο, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί ε, την προσοχή μας ε, και τις ε, ενέργειές μας. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οφείλουν να συνεχίσουν ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων και είμαι σίγουρος ότι τελικά ε, θα μειωθεί αυτή η κατάσταση του λαθρομπορίου τσιγάρων. Θα περιοριστεί. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, και τώρα ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κέσλα ε, κατά πόσον θέλει να τοποθετηθεί σε αυτά που ελέγχθησαν ή μήπω θέλει να τοποθετηθεί αργότερα στις 15 Οκτωβρίου όταν θα έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδα ότι με έχετε καλέσει για τις 15 του μήνα. Θα αξιοποιήσω εκείνη την ευκαιρία για να τοποθετηθώ εκτός και αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις στις οποίες μπορώ να προσπαθήσω να απαντήσω. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ απολύτω με αυτά που είπε ο κύριος Επίτροπος και αν μου δίνετε το λόγο, το μόνο που θα έκανα ήταν να τα επαναλάβω. Ευχαριστώ κύριε Κέσλερ. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανεξαρτησία ε, της Όλαφ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν έχει ζητήσει κανένα άλλο το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά κύριε Επίτροπε για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Τη χαιρετίζουμε και εμείς ε, ως επί τη αρμόδια επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξουμε τις ε, προτάσεις σας, γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα θέματα. Χαιρόμαστε ε, για την συνέχιση της ε, συζήτησης και ελπίζουμε γενικά να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα τόσο όσον αφορά στα θέματα της επικουρικότητας, όσο και στην αναγκαία βελτίωση των διαδικασιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ja, ich fahre dann fort in der Προχωρούμε με την ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο, σημείο 8. Το πρόγραμμα Ηρακλής 3, Ερκούλ 3. Εδώ έχουμε την εισηγήτρια, την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα. Θα ήθελα να την καλέσω λοιπόν να λάβει άμεσα το λόγο και να μας παρουσιάσει την έκθεσή της, το σχέδιο έκθεσης. Συγχωρείτε. Παρακαλώ κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια των προηγούμενων συζητήσεων που είχαμε διεξαγάγει, αλλά και εν ώψη της ε, οικονομικής κρίσης η οποία υπάρχει και συνεχίζεται και των αρνητικών συνέπειών της, έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα το λαθρεμπόριο ή την παρα, αγαθών. Υπάρχουν εθνικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην καταπολέμηση των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων. Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα Ηρακλής 3 ε, ιδρύθηκε το 2004 και στόχος του είναι η προώθηση ε, τέτοιων δραστηριοτήτων προς ε, το τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 2003 το πρόγραμμα αυτό θα λήξει και πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θωρακίσουμε το επόμενο, το πλαίσιο για την συνέχεια του προγράμματος Ηρακλής 3. Πιστεύω πως αναγκαίο είναι να παρέχουμε ε, ως, τους αναγκαίους πόρους για το Ηρακλής 3 όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αυτές οι δραστηριότητες θα ωφελήσουν όλων μας. Θα σας σκεγγραφίσω τώρα τα αποτελέσματα των συζητήσεων που είχαμε σε αυτήν την Επιτροπή αλλά και κατά την παρουσίαση των δύο εγγράφων εργασίας και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, με τους εμπειρογνώμονες ε, και της ε, ακρόασης που διοργανώσαμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Προτείνω 22 τροπολογίες συνολικά οι οποίες έχουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, δηλαδή τον συντονισμό, την διαφάνεια, τα αποτελέσματα και τη συγχρηματοδότηση. Και πολύ σύντομα θα ήθελα να σχολιάσω το την κάθε μία από αυτές τις κατευθύνσεις. Καταρχάς τον συντονισμό. Πιστεύω πως πρέπει να διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό σε τρία επίπεδα. Καταρχάς μέσα στις διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και τέλος στα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Οι τροπολογίες που καλύπτουν αυτόν τον τομέα είναι οι 2, 5 και 7. Και είναι σημαντικό αυτό, πιστεύω, ε, διότι με μία αποδοτική διακρατική συνεργασία μπορούμε να καταπολεμήσουμε το, το λαθρεμπόριο. Μας, ε, έχουμε μία έλλειψη πληροφοριών και αυτή η έλλειψη πληροφοριών μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα όπως οι ε, αλληλοεπικαλύψεις. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που παρέχουν χρηματοδότηση και τεχνολογική και τεχνική βοήθεια, την Digitex για παράδειγμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και, αποδοτικότερη, και αποδοτικότερο συντονισμό στις υπηρεσίες που παρέχονται. Το δεύτερο ερώτημα, το ερώτημα της διαφάνειας. Πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε καλύτερα βελτιωμένα μέτρα για την βελτίωση της διαφάνειας και προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρέχει κάθε χρόνο σε εμάς στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο την, ε, το state of play, την ισχύουσα κατάσταση εφαρμογής του προγράμματος και τα δεδομένα όσον αφορά την χρηματοδότηση, αλλά και στοιχεία για, το, για τις αλληλοπικαλύψεις με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό φυσικά πρέπει να, είναι, να γίνεται με τρόπο καθόλου αδιάφανο και άμεσα προσβάσιμο σε όποιον επιθυμεί να λάβει πληροφορίες. Οι τροπολογίες 12, 16 και 17 ασχολούνται με αυτό. Τρίτος τομέας, τα αποτελέσματα. Αυτό το τομέα ήταν αντικείμενο συζητήσεων σε όλες τις ε, σχετικές εκθέσεις τις οποίες ε, με τις οποίες ασχολούμαστε εδώ στην Επιτροπή. Εγώ προτείνω η Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες ε, απόδοσης και να τους συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, διότι αυτοί οι δείκτες, αυτά τα εργαλεία θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος αυτού επευκαιρία αυτή προτείνω να μεταφέρουμε τους στόχους από το παράρτημα του κανονισμού κατευθείαν στο, στο κυρίως κείμενο του κανονισμού, του κανονισμού. Οι σχετικές τροπολογίες είναι οι 4, 8 και 9. Τέλος, το ζήτημα της συγχρηματοδότησης. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης ακούσαμε ότι ορισμένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη εξέφρασαν ανησυχία για το επίπεδο της συγχρηματοδότησης. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθούν τα επίπεδα συγχρηματοδότησης στο 80% σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη που ε, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Φυσικά ταυτόχρονα διατηρώντας μεγάλη διαφάνεια σχετικά με το πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη. Έχω κάποια ερωτήματα αναπάντητα και θα ήθελα αυτά να απαντηθούν πριν καταθέσω σχετικές τροπολογίες για τον τομέα αυτών της συγχρηματοδότησης και θα ήθελα επευκαιρία να καλωσορίσω από τη... ξανά τον κύριο Κέσλερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και χαίρομαι επίσης και για την συνεργασία που είχαμε με το επιτελείο σας. Ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω αυτά τα ερωτήματα και να ακούσω τι έχετε να πείτε για τον στόχο. Ποιος είναι ο γενικός στόχος της ε, Όλαφ και με ποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε να επιτύχετε την βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη μεταξύ τους και στις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις αλληλοεπικαλύψεις ε, από τις ε, διάφορες γενικές διευθύνσεις. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να ακούσω την γνώμη σας είναι το κενό της χρηματοδότησης που παρατηρείτε. Η συμφωνία PMI εκπνέει το 2016 και θα με ενδιαφέρε πολύ να μάθω την συνέχεια την οποία οραματίζεστε. Πώς θα χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμα μετά το 2016. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα ένα τελευταίο σχόλιο. Αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μία πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πάνω στην διαχείριση του προγράμματος, όντας ε, ταυτόχρονα διαχειριστής του προγράμματος και ελεκτής της ε, σωστής εφαρμογής του. Εσείς πιστεύετε πως υπάρχει όντως σύγκρουση συμφερόντων, όπως εξεφράσε το ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ε, ήθελα απλά να σας δώσω το λόγο. Μπερδεύτηκα γιατί η κυρία προηγουμένως ε, προείδρευε και μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Δεν έπρεπε να λάβω λόγο χωρίς να μου το δώσετε. Λοιπόν, ε, θα απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις ε, και μετά θα δώσω το λόγο στον αρμόδιο για το πρόγραμμα Ηρακλής. Όσον αφορά την σύγκρουση συμφερόντων, κοιτάξτε, ε, πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό. Η Όλαφ ε, Επίσης, ε, είναι Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάγεται ή έχει αρμοδιότητες χάραξης πολιτική, συμβάλλει στην εκπόνηση νομοθεσίας, στον ίδιο πάλι τομέα ε, με, τα, με δύο άλλα προγράμματα, το, με τα δύο αυτά προγράμματα, το Περικλής και το Ηρακλής, με τα δύο λοιπόν αυτά προγράμματα, επιδιώκει τους ε, ίδιους στόχους ε, που είναι αρκετά περιορισμένα ε, κάτω από το ευρύ, κλίμα, πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντως εντάσσονται και αυτά σε αυτό τον τομέα, σε αυτό το πεδίο. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις ερευνητικές ε, αρμοδιότητες και της Όλαφ και τις αρμοδιότητες που έχει για χάραξη πολιτικής. Όμως εδώ πρόκειται για δύο ε, διαφορετικές λειτουργίες της ε, Όλαφ και η επιλογή πολιτική κατά της απάτης, ε, ερευνητική πολιτική, όλα αυτά στον ε, ένα και μόνο φορέα, αλλά αυτό είναι, αυτό είναι μια μοναδική περίπτωση χωρίς προηγούμενο που είναι όμως αποτελεσματική, διότι η ε, αρμοδιότητά μας χάραξη πολιτικής απορρέει από τις αρμοδιότητες έρευνας, ερευνών, ελέγχων. Και έτσι λοιπόν προκύπτει και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων Ηρακλής και Περικλής. Εμείς έχουμε καλύτερη κατανόηση του τι πρέπει να χρηματοδοτηθεί γιατί έχουμε τέτοιου είδους ε, εμπειρία. Και νομίζω ότι εμείς γνωρίζουμε πώς μπορούν να, ε, να τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ε, παρεπιπτόντως τα προγράμματα αυτά τα χρησιμοποιούμε εμείς αλλά τα ζητάμε εμείς αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς που σημαίνει ότι δεν εποφελούμεθα από αυτά τα κονδύλια αυτά ε, διοχετεύονται απευθεία στα κράτη-μέλη άρα δηλαδή και κάτω από αυτό το πρίσμα δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων Κατόπιν, όσον αφορά, δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει στις ερωτήσεις σας, αλλά αναφερθήκατε στο θέμα του ποσοστού χρηματοδότησης. Ζητώ από εσάς ως ε, Κοινοβούλιο να στηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος το πρόγραμμα αυτό να μην επιτύχει τους στόχους του. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που αντιτίθενται σε υψηλά ποσοστά χρηματοδότηση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι επίση αλήθεια ότι ορισμένε ε, δαπάνε ε, είναι αρκετά υψηλέ. Δόθηκαν, α πούμε, ένα-δύο εκατομμύρια για ένα και μόνο σκάνερ. Όμω ο σκάνερ είναι σημαντικό για να αποφεύγεται το λαθρεμπόριο. Και αυτό το χρειάστηκε, αυτό το σκάνερ το χρειάστηκε ένα κράτο μέλο, αλλά αυτό είναι και το πιο εκτεθειμένο που φέρει το μεγαλύτερο βάρος ε, του αγώνα ε, κατά του λατρεμπορίου. Ε, αυτό λοιπόν το κράτος μέλος είναι πιο εκτεθειμένο, έχει πιο πολλές δαπάνες ε, και κάνει τη δουλειά με μεγάλη δέσμευση, η οποία μας δουλειά αυτή αποβαίνει προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κράτος μέλος να πληρώσει εκατομμύρια για ένα ή για κάποιο σκάνερ και αν το ποσοστό χρηματοδότηση είναι πολύ χαμηλό, καταλαβαίνετε ότι ε, δεν θα ε, εφαρμοσούν αυτά τα προγράμματα. Άρα πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα, ε, όσον αφορά στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ε, ε, πράγματι θα χρηματοδοτηθεί από τον γενικότερο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρε και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες εμείς εδώ είμαστε. Συνάδελφό μου σας δώσω πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέσλερ. Συνάδελφοι Γιούγκ και Μπαλτσίτη θέλουν το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ντε πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά. Είναι ένα σχέδιο αυτό που περιλαμβάνει πάρα πολλές συστάσεις. Ως προς τη χρηματοδότηση όμως δεν άκουσα την, την απάντηση αν η Φίλιπ Μόρις εξαφανιστεί ως εταίρος μας σε αυτή τη συμφωνία, από πού θα βρούμε χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλο το ποσό, 10 εκατομμύρια αν δεν απατώμε. Αυτό θα έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να το συμπληρώσει αυτό με κάποια μέσα ε, κοινοτική δωρεάς. Από εκεί και πέρα το έγγραφο εργασίας έχει πολύ λεπτομερείς πληροφορίες. Η Γενική Διεύθυνση Ταξίδι, ΟΛΑΦ, η ΖΕΟΜΕΔ. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται και στο οποίο δεν έχω καταφέρει να απαντήσω ακόμα είναι το εξής. Γιατί η Γενική Διεύθυνση Ταξίδι δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η ΟΛΑΦ, δηλαδή ε, παρόλο που δεν μπορούμε να έχουμε σαφή απάντηση σε όλα αυτά, είναι κάπως περίεργο αυτά να γίνονται παράλληλα. Άλλωστε τα χαρτιά αυτά δεν ήταν ποτέ αποτελεσματικά. Όταν έχουμε λοιπόν αντιθέσεις στο εσωτερικό της Επιτροπής, πώς μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι με αποτελεσματικό τρόπο. Και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι και το εξής. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρίσιμα στοιχεία για τις επιδόσεις των κρατών μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να γνωρίζουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα που βρίσκονται στο δημόσιο κορβανά. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση της Όλαφ. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα κείμενο που να τα διευκρινίζει κάπως όλα αυτά ο έλεγχος του προϋπολογισμού δεν είναι εφικτός παρά μόνο όταν ε, κάποιες πληροφορίες είναι ε, σωστά διαθέσιμες. Εάν η Επιτροπή κρατά πληροφορίες για τον εαυτό της με εμπιστευτικό τρόπο, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχουμε τους δείκτες για την ασφάλεια των ε, επιδόσεων και γνωρίζουμε και το λόγο ύπαρξή τους, ύπαρξής ο αριθμός των κατασχέσεων, ο αριθμός των δεσμεύσεων. Αυτό, με αυτό αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ή πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία των ε, μέτρων που λαμβάνονται. Άλλο, άλλη ένδειξη, άλλος δείκτης ε, μπορεί να είναι πιο χρήσιμος. Να έχουμε το κριτήριο της ενημέρωσης, των συσκέψεων, των συναντήσεων για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσοι έχουν συμμετάσχει, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και ποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί. Πράγματι βελτιώνονται τα πράγματα στην πράξη. Με όλες αυτές τις συνεδριάσεις και τις συσκέψεις ε, έχουμε ε, προστιθέμενη αξία. Και δεν το λέω για να ε, επικρίνω τα πιο ευπαθή κράτη-μέλη, τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν υπερβολικό ένα κράτος μέλος που είναι πιο ευπαθές θα, λέγα, θα λέγαμε σήμερα, ενδεχομένως αύριο να μην είναι, κάποια άλλα να μπουν στη θέση του. Θα προτείνω λοιπόν και προτιμώ βεβαίως να προβλέψουμε απαραίτητες εξαιρέσεις, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις Δηλαδή μια εξαιρετική περίπτωση δεν μπορεί να είναι ένα κράτος το οποίο παγίως θεωρείται ως ευπαθές κράτος και άρα εκτίθεται βεβαίως σε μεγαλύτερο ποσοστό σε τέτοιου είδους λαθρεμπόριο. Πολύ λοιπόν μια σειρά ερωτήσεων ε, και επόμενος ο κ. Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να, πω, να απευθυνθώ προς την εισηγήτρια και να πω ότι έχει συντάξει μια πολύ ποιοτική έκθεση, παρόλο που είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μάθαμε πολλά για την ανεξαρτησία της Όλαφ. Και αυτό το ζήτημα το θέσαμε κατά μέρος όταν συζητήσαμε τις μεταρρυθμίσεις για την Όλαφ. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε το κείμενο που έχουμε. Είναι ανεξάρτητο όργανο η Όλαφ, αλλά α, είναι μέρος, αποτελεί μέρος της διάρθρωσης της διοικητικής δομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα ζήτημα που έχει αναφερθεί το 2011 επίσης. Και ε, αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με την ανάκτηση πόρων κονδυλίων που δεν έχουν αξιοποιηθεί ε, ορθά στα κράτη-μέλη. Έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, απολύτως ξεκάθαροι. Και θα πρέπει να το γράψουμε επί χάρτου, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση των παρανόμως χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, γιατί αλλιώς εγείρεται ζήτημα ευθυνών. Ο κύριος Κέσλερ έχει ήδη δηλώσει με πολύ διπλωματικό τρόπο ότι η Όλαφ σήμερα ε, ασκεί καθήκοντα τα οποία τυπικά δεν τις αναλογούν. Ενδεχομένως με αυτή την νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημοσίου Κατηγόρου, ε, το EPPO, ε, το πρόβλημα αυτό θα εξαφανιστεί αλλά ως προς την ανάκτηση παρανόμως χρησιμοποιηθέντων πόρων ή κονδυλίων ή πιστώσεων, αυτό είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατσίτης. Ο κύριος Γκάια. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο αυτό της έκθεσης ε, που ε, εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Ε, με τα περισσότερα από αυτά που είπατε ε, συμφωνώ. Όμως ε, για μένα υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι μεγάλη σημασία και που θα ήθελα να συζητήσω με σας και τους συναδέλφους σας. Και εδώ συμφωνώ με αυτό που ο Ντεγιόν σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, Υπάρχει ένα κοινό καθήκον για την Κομισιόν, για τα κράτη-μέλη, που είναι να προστατεύουν τα όρια, να εμποδίζουν το λαθρεμπόριο και με τον τρόπο αυτό να ε, προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή αυτό καθιστά απαραίτητο να υπάρχει συγχρηματοδότηση. Κατανοώ αυτό που λέτε ότι υπάρχουν κρατημέλη και προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρηματολόγησε και ο κύριος Κέσλα ότι υπάρχουν κρατημέλη που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όμως ε, δεν έχει νόημα ευθύς εξ αρχής να επιλέξουμε ορισμένα κρατημέλη τα οποία να απαλλάσσουμε σε κάποιο βαθμό από τα καθήκοντά τους. Γιατί τι θα γίνει τελικά αν ε, με τα ποσά τα οποία ε, καταβάλλονται από την ε, ε, βιομηχανία τσιγάρων δεν έχουμε πια τον έλεγχο, αν χάσουμε τελείως τον έλεγχο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δύσκολο για πολλά κράτη-μέλη να λάβουν τις ευθύνες τους. Κατάλαβα τους χάρη ότι στη Γερμανία υπάρχει ένα συνταγματικό πρόβλημα είναι δύσκολο να γίνει αυτό το περίφημο earmarking. Από την άλλη όμως ε, τα κράτη-μέλη έχουν λάβει τεράστια ποσά ακριβώς για να εκπληρώνουν αυτά τα καθήκοντα. Άρα δηλαδή αυτή τη σχέση θα ήθελα να την συζητήσουμε λίγο πιο ευέλικτα. Και όχι απλά να πούμε ότι εντάξει ξέρετε ε, θα επιλέξουμε έναν αριθμό ε, κρατών μελών ε, και εκεί θα είναι υψηλότερη η συγχρηματοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί στην περίπτωση αυτή ε, θα έρθουν κράτη-μέλη ή όλα τα κράτη-μέλη ε, θα μας καταθέτουν τον λογαριασμό, θα λένε εμείς ε, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας, παρακαλώ ελάτε χρηματοδοτήστε. Σίγουρα δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ένα Ηράκλειο έργο. Όμως συμφωνώ με τον συνάλφο Ντιό ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Και το άλλο που θέλω να πω αφορά στον όγκο. Κοιτάξτε, με ε, ξέπληξε λιγάκι το γεγονός ότι στα μέτρα αυτά προστασίας των συνόρων η Κομισιόν ε, εστιάζει την προσοχή της κυρίως στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν λέω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά κοιτάξτε, οι εκθέσεις της Europol δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόνο αυτός. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ε, οντί λατρεμπορίου ε, εισαγωγή λατρέων τσιγάρων στην Ευρώπη και η Ανατολική Ευρώπη αυτό είναι μόνο ένας, μία οδός. Ο κύριος ε, Σεμέτα είπε ότι αυτό θα ληφθεί δεόντως υπόψη και είναι αρκετά χρονοβόρο το θέμα, μόνο που τι το ερώτημα τι θα γίνει με το πρόγραμμα και τι θα γίνει και με τα κράτη-μέλη, τα οποία χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη. Σε αυτά λοιπόν τα δύο θέματα, έκταση του προγράμματος και κράτη-μέλη για τα οποία, ε, τα οποία ε, πρέπει να ε, βοηθηθούν από το πρόγραμμα Ηρακλής 3. Επόμενος ο κύριος Σκυλακάκης. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια γιατί πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση και έχω να κάνω μόνο μία-δύο παρατηρήσεις. Ξεκινάω λοιπόν από αυτά. Όσον αφορά τα ε, τροτά κράτη-μέλη, εγώ έρχομαι από ένα τέτοιο, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι λάθος να χορηγούμε αυτές τις εξαιρέσεις. Γιατί όσο Όσο αυξημένο είναι το ποσοστό της συγχρηματοδότησης, τόσο περισσότερο ενδίδουν τα κράτη-μέλη στον πειρασμό να προβαίνουν σε κακοδιαχείριση. Όταν έχουν το 90% συγχρηματοδότηση προγραμμάτων, ε, κατά κάποιον τρόπο εξωθούνται στο να τα δαπανούν ε, λανθασμένα. Αν θέλει κανείς πραγματικά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το λατρεμπόριο τσιγάρων, τότε πρέπει να γνωρίζει ότι το κέρδος είναι πολλαπλάσιο αυτού που επενδύεται για την αντιμετώπιση του λατρεμπορίου. Άρα δηλαδή καταλήγω στο ότι να μην χορηγούμε εξαιρέσεις, να μην εξαιρούμε κράτη-μέλη σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο που θέλω να θίξω αφορά στις, ε, στους επιτόπιους ελέγχους από πλευράς Όλαφ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Όλαφ να κάνει ε, στην περίπτωση αυτή ελέγχους μετά από δική της πρωτοβουλία. Γνωρίζουμε από ε, δείκτες της ε, Transparency International από τούτου φορέα και αναφέρομαι στους δείκτες που έχουν σχέση με το δημόσιο τομέα και με την δωροδοκία σε συγκεκριμένους δημόσιους οργανισμούς. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι σε ορισμένα κρατημέλη υπάρχει εκτεταμένο φαινόμενο δωροδοκίας στα τελωνία. Κυρίως ε, όταν ε, οι οδοί, οι αποστάσεις, μάλλον οι οδοί είναι μεγάλες, ε, αυτές που διανύουν οι λατρέμποροι. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφθορά γίνεται συστημική. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, βρει κανείς κάποιον που θα είναι πρόθυμος να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες περί διαφθοράς. Άρα δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι πρέπει μόνη της να επεμβαίνει η Όλαφ. Σήμερα δεν το κάνει. Οι περισσότερες από τις έρευνες που διεξάγει η Όλαφ ε, προέρχονται από, κάποιες, από κάποιους πληροφοριοδότες. Και τέλος, Όσον αφορά στους δείκτες, χαίρομαι πάρα πολύ που η συγγήτρια υπογραμμίζει ότι οι δείκτες μπορούν να βοηθήσουν γιατί έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, να μην τα χάνουμε, αλλά κυρίως για τα ευάλωτα αυτά τα κονδύλια κατ' ουσίαν λείπουν από ανθρώπους συνταξιούχους χαμηλόμισθους ε, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να περικόπτονται. Συμπέρασμα, πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Ja, Dank, Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε κύριε Σκυλακάκη. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Κύριε Γενικέ ε, Διευθυντά, εμάς μας ανησυχεί η κατάσταση, κυρίως όταν δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με τα χρήματα. Δηλαδή, ε, θα μας ενδιαφέρει να έχουμε εκθέσεις, γιατί όποιος ε, παίρνει χρήματα πρέπει και να ε, μπορεί να ελέγχει τι γίνεται μετά από δύο χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα αν δεν γνωρίζουμε μακροπρόθεσμα τι γίνεται με τα χρήματά μας. Και θα ήθελα να έχω και την δική σας την ε, προσωπική αξιολόγηση για τα χρήματα τα οποία έχουν εισπραχτεί από τις ε, πολυεθνικές ε, τσιγάρων. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια το ύψος των κονδυλίων το διαπραγματεύτηκαν οι Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και αν μπορεί κανείς να απευθύνει μια κατηγορία στην ε, Κομισιόν ε, είναι ότι ήταν πολύ κακή η διαπραγματεύση. 10% πήρε αυτή και 90% τα κρατημέλη και τώρα είμαστε εμείς εκείνοι που καλούμε να υλοποιήσουμε μία σειρά από μέτρα. Άρα δηλαδή ε, πώς εκτιμάτε εσείς τι δυνατότητες έχουμε να αναδιαπραγματευτούμε το θέμα της αποζημίωσης. Εγώ λέω ότι μάλλον δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εσείς έχετε την ίδια άποψη. Και μετά, ε, η Όλαφ έχει έναν κατάλογο του τι πρέπει να γίνει και τι δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια και δεν το έπραξαν. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, μια ολόκληρη σειρά θεμάτων. Ε, κύριε Κέσλερ, ε, κύριε Γενική Διευθυντά, ε, ίσως μπορείτε εσείς ή και οι συνεργάτες σας να τοποθετηθούν. Παρακαλώ. Yes. Uh, I pick four questions Λοιπόν, να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Φίλιπ Μόρις και γενικά οι πληρωμές από την βιομηχανία καπνού και τσιγάρων. Παρακαλώ να μην συγχαίουμε τα θέματα. Καταρχάς θέλω να πω αυτό. Με χαρά απαντώ στις ερωτήσεις και με χαρά θα σας δώσω και όλες τις πληροφορίες. Αλλά αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με τον Ηρακλή 3. Το Hercule 3 δεν έχει τίποτα να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα που έρχονται από τη Philip Morris ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ε, παραγωγής ε, προϊόντων καπνού και τσιγάρων. Ο Ηρακλής είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καπνοβιομηχανία, η μέρος αυτής, είχε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα πριν από αρκετά χρόνια μετά από ε, μια δίκη στη Νέα Υόρκη ε, είχαν λοιπόν φτάσει αυτά τα συμβαλόμενα μέρη σε μια συμφωνία πολύ περίπλοκη και επί τη βάση αυτής της συμφωνίας πληρώνονται ετησίως ποσά από την Φίλιπ Μόρι στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 9,7% των πληρωμών που ε, ε, έγιναν αντικείμενο συμφωνίας επί τη βάση ε, της ε, απόφασης ε, του δικαστηρίου. Δηλαδή 9,7% των ετησίων πληρωμών τους πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο στα κράτη-μέλη. Και πηγαίνει αυτό το 9,7% στο γενικό προϋπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτω από την επικεφαλίδα εισοδήματα, έσοδα μάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πηγαίνει, δεν χαρακτηρίζεται και μαρκάρεται για τον πρόγραμμα Ηρακλής ή για την Όλαφ ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτω από την, ε, τον τίτλο, την επικεφαλίδα «Γενικά έσοδα». Υπ' αυτή την έννοια δεν μας πληρώνει σε καμία περίπτωση ε, η ε, καπνοβιομηχανία. Τα χρήματα που πληρώνει πηγαίνουν στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, τα κονδύλια που πάνε στην Όλαφ πώς αξιοποιούνται, ε, πώς δαπανώνται από τα κράτη-μέλη. Δεν δίνουμε χρήματα απλά έτσι όπως να είναι. Δίνουμε χρήματα βάσει συγκεκριμένων project. Και τρία προγράμματα ή σχέδια είναι επιλέξιμα βάσει του Ηρακλή. Το, πιο, το πρώτο και το πιο ε, ε, και το πιο κονδυλιοβόρο θα έλεγα είναι το πρόγραμμα και το σχέδιο ε, για το τις συσκευές ελέγχου, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης, δηλαδή δορυφόρους, σαρωτές και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολύ εύκολο να ελέγξουμε εμείς κατά πόσο τα κράτη-μέλη τα αγόρασαν πράγματα, τα μηχανήματα και κατά πόσο τα χρησιμοποιούν, γιατί υπάρχουν. Δεύτερο επιλέξιμο σχέδιο και πρόγραμμα, κατάρτιση. Αυτό δεν στοιχίζει και τόσο πολλά. Και τέλος, μικρό μέρος των χρημάτων πηγαίνει στη συνεισφορά προς τα κράτη-μέλη για να μπαίνουν στις βάσεις δεδομένων, να τις συμπληρώνουν, ούτω ώστε να έχουμε επαρκείς βάσεις δεδομένων ε, για να μπορούμε να ανεχνεύουμε το λαθρεμπόριο, την παραποίηση προϊόντων ε, κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι ανοιχτά, δηλαδή διαθέσιμα. Ε, μπορούμε να δούμε πώς οι Όλαφ και τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τα κονδύλια βάσει του προγράμματος Ηρακλής. Ε, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως διαθέσιμες και προσβάσιμες πρέπει να τη ζητήσετε κάθε χρόνο, αλλά και να μην τη ζητήσετε, εμείς κάθε χρόνο συντάσσουμε έκθεση ε, για την αξιοποίηση αυτών των ε, οικονομικών δυνατοτήτων. Για φέτος θα βγει η έκθεσή μας την επόμενη εβδομάδα, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε. Θα την έχετε και αν χρειάζεστε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να μας το ζητήσετε. Αλλά στην έκθεσή μας καλύπτουμε τα πάντα. Επομένως γνωρίζουμε ακριβώς πώς δαπανώνται τα χρήματα από τα κράτη-μέλη, αλλά ε, είναι σαφές, δεν είναι καθόλου απόρριτα τα στοιχεία αυτά, δεν είναι καθόλου ε, εμπιστευτικά. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσουμε την ετήσια έκθεσή μας που θα τα περιλαμβάνει. Στην Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό είδα ότι μια τροπολογία έχει προταθεί ότι δηλαδή δεν θα σας δώσουμε 10 εκατομμύρια π.χ. εάν δεν μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιου είδους στοιχεία σε ένα ασφαλές δωμάτιο και κτλ. κτλ. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος όπως σας λέω να γίνεται κάτι τέτοιο. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια δεν έχουν καμία σχέση με έρευνες ή με οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να, έχετε πρόσβαση σε αυτά. Ε, συν της άλλης, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Γκάιερ. Και εγώ είμαι υπέρ της ευελιξίας. Ήδη έχω αναφερθεί στη δυνατότητα να έχουμε υψηλότερο βαθμό ή υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τέτοιο, ένας τέτοιος αρωτής δεν στοιχίζει ποτέ κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ αν όχι και παραπάνω, 2 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν έναν τέτοιο σαρωτή. Μιλώ βέβαια, αναφέρομαι στους σαρωτές που μπορούν να σαρώσουν ένα ολόκληρο φορτηγό ή ένα ολόκληρο βαγόνι ενός τρένου και εξαιρετικά αποτελεσματικά είναι αυτά τα μηχανήματα για το έλεγχο του λαθρεμπορίου, αλλά είναι και εξαιρετικά ακριβά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε υψηλό βαθμό συγχρηματοδότησης, τα κράτη-μέλη δεν θα τα αγοράσουν ποτέ αυτό το μηχάνημα. Ε, βεβαίως είμαι ευέλικτο και δεν θέλω να πω εκ των προτέρων ποιο κράτος μέλος θα πάρει χ ποσοστό συγχρηματοδότησης και ποιο άλλο κράτος μέλος θα πάρει λιγότερο ή περισσότερο. Διότι βεβαίως πράγματι αλλάζουν τα πράγματα. Σήμερα ε, ε, ε, μπορεί να έχουμε πέντε ευπαθή κράτη και σε έξι μήνες να έχουμε άλλα πέντε. Και συμφωνώ και με τη διάσταση των ανατολικών συνόρων, όπως την ανέφερε ο κύριος Γκάιερ. Ήταν ανατολικών συνόρων η διάσταση αυτή. Στους επόμενους μήνες θα έχουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα ονομάζεται «Ανακοίνωση της Επιτροπής για το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελεία, χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό» διότι πράγματι δεν είναι μόνο τα ανατολικά σύνορα, το φαινόμενο έχει διασπαρθεί ε, γεωγραφικά, κινείται, επεκτείνεται και χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο περιεκτικό, ένα συνολικό σχέδιο. Και γι' αυτό θα έχουμε μια ανακοίνωση γενικότερη για όλη την Ένωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτές τις απαντήσεις που μας δώσατε. Κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να ξαναπάρει το λόγο. Ο κύριος Χέσλιν, παρακαλώ. Η κυρία. Μάλιστα, θα ήθελα να μάθω σε τελική ανάλυση τι γίνεται με τα κονδύλια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε τη λίστα. Την ζητήσαμε, δεν τη λάβαμε. Ε, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αναλάβει ένα έργο και δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Ζητήσαμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα και δεν τα έχουμε λάβει ακόμα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε καλέσει και πολλές φορές εκπροσώπους του Όλαφ. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω άλλη μια φορά, ελπίζω τελευταία, να μας δώσετε τις πληροφορίες που ζητήσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κύριε Κέσλερ, ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, να μας πείτε πότε θα λάβουμε αυτή τη λίστα, αυτό τον κατάλογο. Δεν είμαι βέβαιος. Ε, ε, για ποια λίστα μιλούμε. Έχω ένα γράμμα μπροστά μου, μια επιστολή χωρίς ημερομηνία, την οποία έστειλε ο διευθυντής μου στην κυρία Γκρέσλερ με μια λίστα με τα ποσά που ε, ελήφθησαν από κράτη-μέλη ε, ε, από πλευράς των, ε, της καπτοβιομηχανίας. Για αυτή τη λίστα μιλούμε ή ποιο άλλο κατάλογο χρειάζεται. Κυρία Κέσλερ, ίσως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Ναι, ζητήσαμε να μάθουμε ποια κράτη-μέλη έλαβαν αυτά τα κονδύλια από, την ε, από τις καπνοβιομηχανίες. Και ποια project συγχρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα κονδύλια και σε ποια κράτη-μέλη και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι υποδομές. διότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αυτά τα project δεν λειτουργούν σωστά ή και καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν ανακεφαλαιώνω τι λειτουργεί, εάν λειτουργεί και τέλος ερώτησα εάν η Όλαφ έχει και τελος ρωτησα εαν η κατάλογο που, στον οποίο αναφέρεται η κατάσταση. Επαναλαμβάνω ότι πολλές φορές ζητήσαμε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες και αυτός είναι και ο λόγος μάλιστα που το ζήτησα διότι εμείς χρειάζεται να μάθουμε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα, τώρα έγινε η κυρία Κρέσλε σαφής, κύριε Κέσλερ. Μάλιστα, υπάρχουν τρεις λίστες. που πρέπει να σας δώσουμε από ό,τι καταλαβαίνω η μία, ο ένας κατάλογος είναι ο κατάλογος με τα κονδύλια που έχουν διατεθεί από τις καπνοβιομηχανίες στα κράτη-μέλη σύμφωνα με τις ε, συμφωνίες που έχουν γίνει. Αυτή εστάλη Εάν μας τη ζητήσετε ξανά θα σας την στείλουμε. Η δεύτερη, ο δεύτερος κατάλογος, η έκθεση δηλαδή, αναφέρεται στο πόσα χρήματα έχουν λάβει τα κράτη-μέλη μέσω της Όλαφ από τα κονδύλια του Ηρακλή στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης. Αυτό θα περιέχεται στην έκθεση την οποία όπως κάθε χρόνο καταρτίζουμε για το πρόγραμμα Ηρακλής. Όχι, λάθος, διορθώνεται ο μιλητή. Για πρώτη φορά θα καταρτιστεί λοιπόν αυτή η έκθεση. Την επόμενη εβδομάδα όμω όπως και να έχει θα την λάβετε κυρία Γκρέσλε. Είναι έτοιμη η έκθεση. Την επόμενη εβδομάδα θα την έχετε. Δεν το αποφασίσαμε προχθές αυτό. Έχουμε πάνω από ένα χρόνο που το δρομολογούμε και θα έχετε στη διάθεσή σας την πλήρη έκθεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Και επί τη ευκαιρία, εάν έχετε έτσι αναδρομικά κάποιες ερωτήσεις για τη συγχρηματοδότηση των προηγούμενων ετών πριν το 2011, δεν είναι κάτι το εμπιστευτικό αυτό, δεν είναι απόρριτες πληροφορίες, μπορείτε να τις πάρετε όποτε θέλετε. Τρίτον, αν κατάλαβα καλά, θέλετε έναν κατάλογο του τι δουλεύει και τι όχι κυρίως το ότι δεν δουλεύει στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Ποια είναι τα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Μάλιστα, αυτό είναι μια αξιολόγηση η οποία θέλει χρόνο, αρκετό χρόνο, έτσι ώστε να απαντηθεί σωστά και διεξοδικά, πρέπει να γίνει επιτόπιος, επιτόπια αξιολόγηση σε κάθε κρατός μέλος. Και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, από τις τεχνικές δυνατότητες που έχουν, από την θέληση που έχουν για να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο. Το επεξεργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τις απαντήσεις. Έχω μία ακόμα παρέμβαση από τον συνάδελφο Ντε Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, όπως είδαμε, ε, μεταξύ του κυρίου Κέσλερ και εμού. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν σχετικά με τα 10 εκατομμύρια, τα οποία σύμφωνα και με το λεκτικό συνέδριο λείπουν από το πρόγραμμα λείπουν 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα, παρέχει, θα παρέχουν οι καπνοβιομηχανίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του λαθρεμπόριου τσιγάρων. Καταλαβαίνω ότι όλα λέει ότι αυτό προέρχεται από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι σύπτωση το γεγονό ότι τώρα καταπολεμούμε το λαθρεμπόριο τσιγάρων με ακριβώ τα ίδια χρήματα τα οποία μα διέθεσαν οι καπνοβιομηχανίε. Βλέπω ότι την προσεχή περίοδο κατά τη διάρκεια του προγράμματο Ηρακλή 3 θα έχουμε πρόβλημα, διότι ακόμα λιγότερα κονδύλια θα προέρχονται από, την, από τις καπνοβιομηχανίες. Πιο λιγότερα κονδύλια από αυτά που δαπανούνται για το λαθρεμπόριο καθ' αυτό. Γι' αυτό ίσω εμείς να έπρεπε να ξοδέψουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια για να μάθει και να δούμε εάν το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας ή εάν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας είναι άλλες μορφές λαθρεμπορίου. Η εαν στην κορυφη των προτεραιοτητων μας ειναι άλλε μορφες λαθρεμποριου η φιλιπ για παράδειγμα, διατυπώνει παράπονα για παραποιήσεις προϊόντων της και ίσως θα έπρεπε να αυξήσουμε την χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ιδιαίτερα αν τα κονδύλια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου δεν προέρχονται πλέον από τις καπνοβιομηχανίες. Έπειτα, δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι κυμαίνεται στο ίδιο μικρό σχήματος με αυτό που είπε η συνάδελφός μου κυρία Γκρέσλε. Εγώ θα το προχωρήσω λίγο ακόμα. Ωραία να δώσουμε τους ερωτές αυτούς. Και βασισμένος από την προηγούμενη εμπειρία μπορώ να πω ότι όλοι θέλουν να έχουν τέτοια μηχανήματα. Όλοι. Και οι εκκλησίες θέλουν να έχουν υπολογιστέ και οι τελωνιακοί έλεγχοι θέλουν να έχουν σαρωτές. Όμως, τι κάνει αυτός ο σαρωτής πρέπει να ξέρουμε. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται, ποια είναι τα αποτελέσματα πόσες ε, περιπτώσεις ανάκτησης προϊόντων λαθρεμπορίου έχουν εντοπιστεί χάρη σε αυτούς τους αρωτές. 67,9 εκατομμύρια ευρώ ανακτήθηκαν τον περασμένο χρόνο. Από την άλλη όμως δεν μας λέτε στον στην έκθεση αυτή εάν υπάρχει κάποια σύνδεση στο... ανάμεσα στο πρόγραμμα και σε αυτά τα 67,9 εκατομμύρια. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε τι έχετε δώσει στα κράτη-μέλη και τι αποτέλεσμα είχε αυτό. Και τέλος, πραγματικά πιστεύω ότι ο συντονισμός μέσα στην Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιωθεί, διότι η, διαφθορά είναι, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι κάτι που μας έχετε υποσχεθεί. Μας έχετε δώσει και μια έκθεση για την κατάσταση ε, της διαφθοράς στα κρατημέλη. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω έκθεση. Η έκθεση αυτά είναι διεξοδική και διήρκησε και πολύ καιρό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον... στην ησυχήτριά μας για τα σχόλια. Τέλος, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για σε όλους τους συναντέλφους ε, για τα σχόλιά τους ε, γιατί ήταν ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πολύτιμα και γι' αυτό λοιπόν ε, καλώ όλους τους ε, συγητές σε αμέσως επόμενες ημέρες ε, να συζητήσουν μαζί μου τις απόψεις μας. Και ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους, κυρίως τον κύριο Κέσλα. Και πρέπει να σας πω ότι προσβλέπω στο να έχουμε μια πραγματικά καλή συζήτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους σκιώδεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ε, κλείνει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, και διακόπτουμε τώρα μέχρι αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστούμε. Γεια σας.